Συνάδελφοί μου, καλημέρα σας. Αποφάσεις των συντονιστών στην σε χθες το απόγευμα, 21 Ιανουαρίου. Σα έχουν διανεμηθεί τα αντίγραφα. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει ω τι 12.30, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν. Κύριε Ερτούκ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια αντίρρηση και θέλω να σας την ανακοινώσω. Οι συντονιστές που συμμετείχαν χθες στην συνεδρίασή μας θα αναρωτιούνται για το ότι στο σημείο 4 εμφανίζεται μια ε, απόφαση ότι έχουμε αναβάλει τη συζήτηση του θέματος για την, για του, του πακέτου για την κινητικότητα στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Συζητήσαμε πάρα πολλή ώρα και μάλιστα ε, έγιναν και πολλές αντεγκλήσεις και καταλήξαμε στο ότι υπάρχουν τρεις επιλογές επί των οποίων θέλουμε να ψηφίσουμε. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το αν θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο ή όχι. Ήταν μια ε, χαοτική η, η κατάληξη της συνεδρίασης και πολλοί δεν είχαν ε, καταλάβει τι τελικά συμφωνήσαμε. Αλλά αυτό που σίγουρα δεν συμφωνήσαμε είναι ότι θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Μεταξύ άλλων ε, είπαμε ότι η Πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο Ταγιάννη ώστε να συζητηθεί το θέμα και στη διάσκεψη των Προέδρων και να αποφασιστεί εκεί. Γι' αυτό και θέλω το συγκεκριμένο σημείο της ημέρης της διάταξης να το αμφισβητήσω και ζητώ σήμερα εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών να γίνει ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αρτούκ. Άλλες πρατηρήσεις? Όχι. Κύριε Βαντεγκάμπ, να κρατιέστε. Πρόεδρε, και εγώ ήμουν εδώ στην συνεδρία των συντονιστών χθε το βράδυ. Ήταν πραγματικά μια συνεδρίαση που κανείς δεν κατάλαβε τι έγινε. Δεν ενθυμούμε να λαμβάνουμε τέτοια απόφαση, ούτε κι εγώ. Νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να ξανασυζητήσουμε στις 29 Ιανουαρίου. Άλλοι έχουν σχόλια. Κύριε Τέλιτσκα, και εσείς αν και δεν είστε πολύ καλοξυπνημένος, όπως είπατε νωρίτερα. Πρόεδρε, καλημέρα. Ελπίζω ότι θα με κάνετε να αισθανθώ καλύτερα. Όχι σαν να έχουμε όλες βγει από το τους. Χθες υπήρξε μια σχετική σύγχυση που οφείλεται στις διαφορετικές τοποθετήσεις, φαντάζομαι. Και στο πλαίσιο της Επιτροπής πρέπει να πω ότι οτιδήποτε συζητήσαμε χθες και θα έπρεπε να ψηφιστεί σε ό,τι αφορά το πακέτο κινητικότητας, έδινε αποτέλεσμα 50-50 για τις θέσεις των μεν και των δε. Θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε στο συντονιστέ, αλλά δεν νομίζω να αλλάξει η αναλογία του 50-50. Οπότε νομίζω η ορθή προσέγγιση είναι να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Μεταξύ άλλων είναι και υποχρέωσή μας ως συντονιστών. Εάν δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, χρειαζόμαστε την ε, φωτισμένη καθοδήγηση της Επιτροπής μας. Υπήρξαν τρεις επιλογές που συζητήθηκαν χθε και τους ανέφερε και ένα συνάδελφο προένος λεπτού. Αυτές θα έπρεπε να ψηφίσουμε. Πρόεδρος, δεν ήξερα ότι θα γίνει συζήτηση σήμερα το πρωί. Κύριε Λιμπεράτσκι, εσείς και μετά στην κυρία Νταμάτο. Μισό λεπτό. Ο κύριος Λιμπεράτσκι πρώτος. Ε, έχω ερώτηση. Τι θα έπρεπε να ψηφίσουμε. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα ψηφίσουμε το αποτέλεσμα της συνεδρίας των συντονιστών. Τι ήταν, ήταν αστείο, δεν ήταν αστείο, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θα ψηφίσουμε. Ε. Κυρία Νταμάτο, εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να απαντήσω και στην τελευταία παρέμβαση, εγώ συμφωνώ να ψηφίσουμε όλοι στην Επιτροπή Μεταφορών για τις τρεις επιλογές. Δηλαδή, ή Ολομέλεια, ή στην Επιτροπή, ή Επιστολή στην ΚΟΡΠ. Γιατί οι συντονιστές, ε, στην πλειοψηφία των συντονιστών, δεν βρέθηκε ε, άκρη. Αποφάσισε να σταθμίσει το αποτέλεσμα η γραμματεία, ε, αλλά το λογικό συμπέρασμα αυτή τη στάθμιση είναι να ψηφίσουμε ακριβώ στην ε, πλήρη σύνθεση αυτή τη ίδια τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε κύριε ταμάτο. Τελευταίο. Είναι η τελευταία φορά που δίνω το λόγο. Κύριε Ζλωτόφσκη. Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω καμία αντίρρηση να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Τραν. Καταλαβαίνω όμως ότι θα χρειαστεί και χρόνος για να προετοιμαστούμε για την ψηφοφορία. Εάν αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ευθύ αμέσω, δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ νόημα. Θα έλεγα λοιπόν εντάξει να ψηφίσουμε, αλλά όχι πριν τι 29 Ιανουαρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε. Να θυμίσω τι συνέβη χθες. Χθες στην συντονιστική μας συνεδρίαση σε σχέση με το πακέτο κινητικότητας έθεσε επιτάπητος τρεις εναλλακτικέ που τις ανέφερα μόλις τώρα οι συντονιστέ μας. Πρώτη, ε, ξανά συζητάμε το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών. Δεύτερη, πάμε απευθεία στην Ολομέλεια. Τρίτη, βλέπουμε στην Ολομέλεια τι συνέβη. Η πρώτη επιλογή πήρε 24 ψήφους. Η δεύτερη, να πάμε στην Ολομέλεια, επίσης 24 ψήφους. Η τρίτη επιλογή, που θα ήταν δική μου ευθύνη, ήταν να ζητήσουμε από την Ολομέλεια να προβλέψει στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό, ώστε η Ολομέλεια τελικά να λάβει την τελική απόφαση. Αυτές ήταν επιλογές. Τώρα που μου ζητάτε να ψηφίσουμε σήμερα το πρωί, βρίσκω προσωπικώς δω ότι δεν έχει νόημα, διότι ουσιαστικά καταστά, καθιστά κενές νοήματος τις αποφάσεις των συντονιστών. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξαναψηφίσουμε για να πάμε στην Ολομέλεια ή ε, να ξανάρθει το θέμα στην Επιτροπή Μεταφορών δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία. Και τρίτο, σε αντίθεση με τον κύριο Ρικέ, που με περνάει για την κυρία Μέη, ε, να πω και το εξή. Ότι ε, για αυτό το πακέτο της κινητικότητας κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβουμε και τις ευθύνες μας, έτσι. Έχει κρατήσει πάρα πολύ όλη η συζήτηση. Το θέμα δεν είναι απλώς να αποφασίσουμε τι θα γίνει με την ψηφοφορία. Το θέμα είναι εάν θα αποστείλουμε επιστολή. προς την Ολομέλεια, στην ε, διάσκεψη δηλαδή των Προέδρων, ώστε να αποφασίσουν εκείνοι. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Κυρία Μάισνερ. Ε, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας κανόνος, κανόνας. Με κάθε σεβασμό είπατε ότι αυτό δεν γίνεται. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πρέπει στους κανόνες να καθορίζεται τι ακριβώς επιτρέπεται και τι όχι. Είναι μπερδεμένη η περίπτωση αυτή, δεν λέω αλλά νομίζω ότι έχουμε περάσει ήδη αρκετό χρόνο στη διαδικασία τη λήψη απόφαση. Και το θέμα που μα απασχολεί είναι αν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει εντό αυτή τη θητεία. Το Συμβούλιο έχει ολοκληρώσει τη δική του θέση και γι' αυτό θα έπρεπε να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατό για να δούμε ποια είναι τελικά η πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή μα. Και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συνάδει με του κανόνε, του ισχύοντε. Όπω είπε και ο Ισμαϊ αν οι συντονιστέ δεν μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένη θέση, τότε πρέπει να ρωτήσουμε την Ολομέλεια. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το θέμα, ακόμη και αν δεν είμαστε εισηγητέ ή σκιώδει, που κάτι τέτοιο ε, είναι εφικτό. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουν σαφή εικόνα για αυτό το πακέτο τη κινητικότητας. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε εφορία ακόμα και σήμερα. Κύριε Ταλούντε, έχετε ζητήσει και εσεί το λόγο. την χθεσινή συζήτηση είχαμε τι τρει επιλογέ. Πρώτη, να ξαναπάμε στην Επιτροπή, μετά να πάμε στην Ολομέλεια και τρίτον, να αποστείλουμε επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων. Για να τοποθετηθούν εκείνοι για την όλη υπόθεση. Η δική μου αποψή είναι ότι θα είναι περίεργο να ξανάρθουμε στην Επιτροπή και να ξαναψηφίσουμε την ίδια πρόταση. Εάν ψηφίσουμε στην Επιτροπή, ε, καλό θα ήταν να δοθεί χρόνο για να δούμε τι συμβαστικέ προτάσει και να δούμε τι αλλαγέ μπορούμε να επιφέρουμε ή ενδεχομένω να διατυπώσουμε νέε. Το να πάμε στην Ολομέλεια χωρί να έχουμε συμβαστικέ προτάσει σημαίνει ότι θα υποβληθούν πάρα πολλέ τροπολογίε και πάλι θα προκύψει μεγάλη σύγχυση. Θα είναι περίπλοκη όλη η ψηφοφορία και τα πράγματα θα είναι μπερδεμένα. Οπότε νομίζω ότι απλώ πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στη διεύθυνση των Προέδρων και να πούμε ότι είμαστε ανίκανοι να καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Κοχ και στον κύριο Λιμπεράτσκε Και μετά θα κλείσω η συζήτηση. Ευχαριστώ. Εκτό όσων καταλαβαίνω, είχαμε συμφανίσει είχαμε συμφωνήσει ότι δεν μπορούν να ε, αποφασίσουν επί της διαδικασίας τρίτη, ούτε η νομική υπηρεσία, ούτε η διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό σημαίνει ότι η βάση, τα μέλη της Επιτροπής μας είναι εκείνα που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα πάμε στην Ολομέλεια ή αν θα προκρίνουμε τις δύο άλλες επιλογές. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ε, ότι πρέπει να αποφασίσουμε είτε τώρα να πούμε ότι δεν προλαβαίνουμε ε, σε αυτή τη θητεία να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο φάκελο ή να πούμε με δύο λόγια ότι το αφήνουμε απευθείας για το επόμενο κοινοβούλιο. Κύριε Λιμπεράτσι και μετά να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο κύριος Κοχ έχει δίκιο αλλά θα ήθελα και την άποψη της νομικής υπηρεσίας για την ελευθερία επιλογής που έχουμε βάσει των κανόνων τι ισχύει και τι είναι αντίθετο με τους κανόνες. Για μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ε, δούμε κατά πόσον ε, ψηφίζουμε, ε, αποφασίζουμε σωστά. Μην ξεχνάμε ότι χθε συζητήθηκε στου συντονιστέ. Πριν από δύο εβδομάδε ψηφίσαμε. Θυμόμαστε και τα αποτελέσματα την ε, ψηφοφορία του περσινού Ιουνίου. Τώρα θα ήθελε επιτέλου να τοποθετηθεί η νομική υπηρεσία και την απόφαση, την τελική απόφαση, να την αναλάβει η Επιτροπή Τραν ε, ω ευθύνη. Ευχαριστώ. Να κλείσει η συζήτηση σε συνεδριάσεις συντονιστών λαμβάνονται αποφάσεις και θεωρούνται ηλυμένε. Πρέπει να γίνονται σεβαστές. Χθε δεν υπήρξε απόφαση. Οπότε ήταν σαφές. Έτσι τοποθετήθηκε η πλειοψηφία. Η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών αναπέμπει μάλλον αποστέλει επιστολή στον κύριο Ταγιάννη ώστε η διάσκεψη των Προέδρων να αποφασίσει. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει ψηφοφορία συγκεκριμένα στην Επιτροπή των Μεταφορών. Τώρα, όσοι θέλουν να πάνε στην Ολομέλεια, μπορούν να πάνε στην Ολομέλεια, να οργανωθούν σε ομάδα και ούτω καθεξής. Χθες ήταν απολύτως σαφές ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία ούτε για τη μία εναλλακτική, ούτε για την άλλη. Δηλαδή, ψηφοφορία στην Επιτροπή ή απευθεία στην Ολομέλεια το θέμα. Άρα, εφ' εξής, ε, το θέμα αυτό θα πάει στην ημερήσια διάταξη τη ε, Διάσκεψης των Προέδρων για να αποφασίσουν αν θα πάνε απευθεία στην Ολομέλεια. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία, διότι χθε, κάποια στιγμή, όταν έπρεπε να ληφθεί απόφαση και δεν ε, σχηματίστηκε κάποια πλειοψηφία, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια τη δημοκρατία. Εγώ δεν έχω τέτοια εξουσιοδότηση. Κύριε Αρτούκ, και είναι τελευταία η παρέμβαση, γιατί έχουμε και ψηφοφορία. Ευχαριστούμε. Λίγο σαν το Μαντούρο ήταν όλα αυτά, αλλά τέλο πάντων. Σε κάθε περίπτωση, όπω ε, το είπατε και πολύ σωστά, και το είπε και ο συνάδελφο Νταλούντε, χθε συζητήσαμε τρει διαφορετικέ εναλλακτικέ. Ξανά το είπατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ότι είχαμε αυτέ τι τρει. Όμω εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ουσιώδου σημασία. Γιατί δεν θα ε, ξεκαθαριστεί στα πρακτικά ότι οι επιλογές ήταν τρεις και το αποτέλεσμα, η έκβαση ήταν ότι θα αποσταλεί επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να παραπέμψει το θέμα στην διάσκεψη των Προέδρων και να αποφασίσουν εκείνοι πώς θα προχωρήσουμε. Πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στα πρακτικά και ασχέτω αυτού, στην Επιτροπή Μεταφορών αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, διαθέσει και συνάδελφοι που θα ήθελαν να αποφασίσουμε επί τη διαδικασία. Δεν μπορεί να λέμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ψηφοφορία. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την Επιτροπή Μεταφορών στο σύνολό τη. Όχι από έναν ή δύο ή τρει συναδέλφου μεταξύ ημών. Κύριε Αρτούγκ θα αλλάξουν τα πρακτικά. Οι τρεις επιλογές θα αναφέρονται ξεκάθαρα. Με την αποστολή από το απόγευμα σήμερα κιόλα προς τον κύριο Ταγιάννη που θα υπογραμμίζει το γεγονός ότι το όλο θέμα ανατίθεται ως ευθύνη στην Ολομέλεια, δηλαδή στην ουσία στη διάθεση των Προέδρων. Τώρα, να μου ζητάτε να ξαναψηφίσουμε για τις τρεις επιλογές εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών δεν είναι δυνατόν. Δεν θα ξανανοίξουμε τη συζήτηση. Δεν είμαι εδώ για να κάνουμε ε, φιλολογική συζήτηση. Το συζητάμε και μετά. Αλλά κάποια στιγμή, όταν πρέπει να ληφθεί απόφαση και δεν προκύπτει πλειοψηφία, δεν προκύπτει πλειοψηφία. Κύριε Τελίτσκα, τελευταία Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει βγει κάποιο συμπέρασμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία. Απόφαση υπάρχει, αλλά ε, αυτά είναι δικά σα συμπεράσματα. Και δεν είμαι βέβαιο αν κάποιο σα στηρίζει ω πλειοψηφία. Καταλαβαίνω, ε, δεν καταλαβαίνω μάλλον γιατί αυτέ τι τρει επιλογέ δεν ψηφίζονται εδώ στην Επιτροπή. Και θα συμφωνήσω με αυτό που ο κύριο Κοκ, ο κύριο Έρτουγκ, ο κύριο Λεμπεράτσκι, η κυρία Νταμάτο. Εμεί ω Επιτροπή Μεταφορών θέλουμε να αποφασίσουμε και μετά να πάει το όλο θέμα στην, ε, στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Δεν καταλαβαίνω απλώ γιατί θα στείλετε μια επιστολή στην διάσκεψη των Πρόεδρων. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Μεταξύ τη συνεδρία των συντονιστών και τη ΚΟΠ υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται Επιτροπή των Μεταφορών. Η Επιτροπή των Μεταφορών δεν μπορεί να επεκδεθεί των ευθυνών τη. Είναι λε και μα λέτε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τι ευθύνε μα με την προσέγγιση σα. Θέλω να το σημειώσετε αυτό. Ευχαριστώ. θα λήξει η συζήτηση και θα πω απλώ το εξή. Σα ε, καταλαβαίνω πολύ καλά, κύριε Τελίτσκα. Το πρόβλημα όμω ουσία ε, χθε και ψηφίσαμε δύο φορέ είναι ότι δεν υπήρξε πλειοψηφία για τη μια λύση ή για την άλλη. Δεν ε, τα βγάζω από το μυαλό μου, εδώ ήσασταν και τα χαρτάκια τα ε, μάζεψε ο κύριο Ράντεκ, έτσι δεν είναι, για να μετρήσει. 24 ήταν υπέρ τη λύση τη Ολομέλεια, 24 τη ε, αποστολή του θέματο στην ε, Επιτροπή μα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία, άρα ολοκληρώνω και κλείνει η συζήτηση. Με συγχωρείτε, αλλά Πρέπει να υπάρχουν κανόνε για αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνε για του συντονιστέ εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία. Ποιοι είναι οι κανόνε, η γραμματεία πρέπει να ξέρει, η Επιτροπή μα έχει δικαιώματα. Θέλουμε να ξέρουμε του κανόνε. Κοιτάξτε, ο κανόνα είναι απλό. Όταν σε συνεδριάσει συντονιστών δεν υπάρχει πλειοψηφία, αν ήταν 25-24 δηλαδή κάτι από τα δύο θα είχε περάσει, τότε λέμε δεν υπάρχει πλειοψηφία. Ο κανόνα λοιπόν είναι ότι το όλο θέμα πηγαίνει στη διάσκεψη των Προέδρων. Η Ολομέλη αποφασίζει.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 Προχωρούμε ευθύ αμέσω με την όλη συζήτηση για τους κοινού κανόνες που εξασφαλίζουν την ε, διασύνδεση του συστήματος αεροναυτιλίας μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της, της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ένωση, έκθεση του κυρίου Τέλιτσκα. Έχουμε και την έκθεση Ζλοτόφσκι και την έκθεση της κυρίας Ντεμόντε. Και τις τρεις αυτές, εκθε... τρεις αυτές εκθέσεις που έχουν να κάνουν με το Brexit σε περίπτωση απουσία συμφωνίας θα τις συζητήσουμε τώρα. Θυμίζω ότι οι συντονιστές ε, ε, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την απλουστευμένη διαδικασία βάσει του άρθρου 50 του ιστορικού κανονισμού. Η διαδικασία θα είναι η εξής είτε θα προχωρήσουμε χωρίς την υποβολή τροπολογιών μετά την ε, σημερινή συζήτηση και σε αυτή την περίπτωση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροποποιήσεις θα πάει απευθεία στην Ολομέλεια. Εκτός εάν προβάλλουν αντίρρηση ένας αριθμός βουλευτών από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που θα εκπροσωπούν το λιγότερο πέντε ε, βουλευτές. Η άλλη δυνατότητα είναι να εγκριθούν τροπολογίες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση μόνον οι ίδιοι εισηγητές μπορούν ε, να υποβάλουν τροπολογίες προτείνοντάς τες στα μέλη της Επιτροπής Τραν. Και αν δεν υπάρξει αντίρρηση ενός ε, ικανού αριθμού βουλευτών ή μιας περισσότερων πολιτικών ομάδων που να φτάνουν τον αριθμό των πέντε, το ξαναλέω πέντε τουλάχιστον βουλευτέ. τότε αυτές οι τροπολογίε θα θεωρηθούν εγκεκριμένε. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσει στις τροπολογίε θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία στην διεξαγωγή της Επιτροπής μας στην επόμενη συνάντηση. Ευθύ αμέσω ο λόγο στον κύριο Τέλιτσκα, που είναι ένα από του εισηγητέ για το θέμα αυτό. Κύριε Τέλιτσκα, έχετε το λόγο. Uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για αυτά τα εισαγωγικά σας λόγια επί της διαδικασίας. Συνάδελφοι, έχουμε πολύ σφιχτό πρόγραμμα και προκειμένου να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να τύχει της πλειοψηφίας και στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι στις συζητήσεις με τους ε, σκιώδεις συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε κοινή στάση μεταξύ των ε, εισηγητών και των σκιωδών έως σήμερα το βράδυ. Έχει προγραμματιστεί και συνεδρίαση των σκιωδών σήμερα και εγώ είμαι διατεθειμένος να αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαστεί. Γιατί το θέμα είναι σημαντικό και έχει σημαντικές επιπτώσεις. Θέλω να τονίσω ότι τα όσα προβλήματα έχουμε μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει δεν οφείλονται σε έλλειψη πρωτοβουλίας από την DG Move. Λαμβάνουμε όμως μία πρόταση αρκετά καθυστερημένα, αργοπορημένα. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες της Κομισιόν ε, θα έπρεπε να είχαν προβλέψει ότι μπορεί και να πηγαίνουμε σε σκληρό Brexit και η απλουστευμένη διαδικασία την οποία αναγκαζόμαστε να πάρουμε οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έγιναν τα πράγματα ε, όπως έπρεπε από την Κομισιόν, όχι από την DigiMove κεντρικά. Το δεύτερο θέλω που θέλω να πω, πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου που χρειάζεται για κάθε ε, κανονισμό, είτε πρόκειται για επίγοντα κανονισμό, είτε όχι. Βλέπουμε εδώ ε, ότι πολλοί ε, συνάδελφοι κάνουν το ίδιο σχόλιο. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Και αυτές δεν είναι σαφές. Δεν υπάρχει μελέτη επιπτώσεων. Και αυτό έχει αναδειχθεί και στις συζητήσεις μας με τους σκιώδεις. Ο κύριος Σελμάιερ ε, μας απάντησε ότι αν επρόκειτο να γίνει ε, μελέτη αντικτύπου θα μας προλάβαινε το ίδιο το Brexit. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική αυτή η απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ε, υπερβαίνει έτσι κι τα όρια των ευθυνών της Digimove. Και θέλω να τονίσω τα εξή. Πρώτον, με κάθε σεβασμό στους Βρετανούς συναδέλφους μου, γνωρίζουμε όλοι ότι οτιδήποτε συμβεί από σήμερα έως το Brexit, ανεξαρτήτως του τι είδους Brexit ε, γίνει τελικά, εκτός αν υπάρχει συμφωνία η οποία θα συναυθεί πριν από το Brexit, αυτό καθε αυτό, θα γίνουν μελλοντικέ διαπραγματεύσει για όλε τι συμφωνίε. Και φυσικά ό,τι κάνουμε τώρα με κάποιο τρόπο διαμορφώνει και τι διαπραγματευτικέ μα θέσει για το μέλλον. Θέλω λοιπόν να πω ότι στη βάση όλων αυτών δεν θα ήθελα να, να πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερες φιλοδοξίες από αυτές που το πεδίο ισχύω ορίζει. Και αυτό δεν το λέω αρνητικά, ούτε θέλω να προκαταλάβω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με την διαπραγματευτική, διαπραγματευτική μας θέση για το μέλλον, αν τέτοια καταρτιστεί. Πάντως, θέλω να πω ότι η διαπραγματευτική μας θέση θα πρέπει να, ένα, ε, ωφελεί τους καταναλωτές, συνδεσιμότητα και τις επιχειρήσεις μας και θέλω να τονίσω και να επισημάνω τα εξή ζητήματα. Γιατί είναι η πρώτη και η μοναδική ευκαιρία που θα έχουμε για να καταρτήσουμε μια έκθεση με την οποία θα ζητούμε διευκρινήσεις από την Κομισιόν. Οπότε πολύ σύντομα θα σας τα πω. Η ίδια η έκθεση είναι ε, σύντομη. Πρώτον, το ερώτημα της, ε, της ε, θέσπισης ανώτατων ορίων, το κάπιν. Θα καταλάβαινα αν αυτή η διάταξη συνδεόταν απευθείας με αυτό που είπα νωρίτερα. Με το σε περίπτωση που αν δεν δηλαδή ορίσουμε ανώτατα όρια, αυτό μπορεί να διαμορφώσει την μελλοντική διαπραγματευτική μας θέση ή την μελλοντική συμφωνία που θα συναυθεί. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί οτιδήποτε αποφασίσουμε εδώ, ε, αν ε, θεσπίσουμε δηλαδή ανώτατα όρια, αυτά τα ανώτατα όρια θα ισχύουν αμοιβαίως. Άρα το αποτέλεσμα θα πρέπει να επιτρέπει τον τάδε αριθμό δικαιωμάτων και συχνοτήτων ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην αγορά. Και όλα αυτά θα σήμαινε ότι θα υπήρχαν συγκεκριμένε επιπτώσεις και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές γιατί πολλά από αυτά έχουν ήδη συμβεί. Πολλοί έχουν για παράδειγμα αεροπορικά εισιτήρια για ταξίδια που θέλουν να κάνουν για παράδειγμα Άρα αυτό έχει και δευτερογενεί επιπτώσει και για του καταναλωτέ και για τι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά και για τι επιχειρήσει συγκεκριμένα στον τουρισμό. Άρα εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά θα μα προκαλέσει μεγάλε δυσκολίε και θα πρέπει να βρούμε ε, μια διέξοδο από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε βρεθεί με τρόπο που δεν θα έχει αρνητικέ επιπτώσει σε κανένα από αυτά τα θέματα. Δεύτερο, και εδώ θα ήθελα πραγματικά διευκρίνηση από την Κομισιόν είναι το ερώτημα της, των δομών ιδιοκτησία. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ δύσκολο ταυτόχρονα. Γιατί έχουμε ήδη λάβει από διάφορα σχόλια από τους συναδέλφους ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις από αυτού του θέματος. Ε, σχετίζεται με την αφετηρία του καθενός, με το τι είδους αεροπορικές εταιρείες υπάρχουν στην κάθε χώρα και ποια είναι τα επιχειρηματικά μοντέλα που υπάρχουν στην κάθε χώρα. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει να είναι κάπου, κάπου στη μέση, μια χρυσή τομή αν θέλετε. Και η σημαντικότερη ανησυχία μου είναι ότι δυστυχώς μας πιέζει τρομερά ο χρόνος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, εισαγάγουμε οποιαδήποτε αναδόμηση οποιασδήποτε εταιρεία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει ε, βεβαίως κανείς να λαμβάνει υπόψη και το επιχειρηματικό μοντέλο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς ε, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί από την Κομισιόν και αυτό, σε αυτό θα κατατείνουν οι προσπάθειές μας το απόγευμα με τους συντονιστές. Το άλλο θέμα ε, που είναι... Για την κατανομή των ποσοστώσεων. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε τις ε, τι ευθύνε που έχουμε, αυτό δεν είναι μόνο ενδοκινοτικό ζήτημα. Κατά κύριο λόγο είναι πράγματι ενδοκινοτικό, αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα. Και τελική παρατήρηση. Έχουμε ορίσει μια ημερομηνία συγκεκριμένη. Όμως, θα πρέπει να εξετάσουμε και την άλλη πρόταση. Θα δούμε ε, για παράδειγμα για τον Οργανισμό για την, για την Ασφάλεια της Αεροπορίας δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Οπότε το ερώτημα εδώ που έχει πολλές διαστάσεις, η βασική διάσταση όπως είναι τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Γιατί εδώ θα υπάρξει ένα θέμα αρμοδιοτήτων. Και όλα αυτά θα ε, έρθουν στο φως και στις μελλοντικές συζητήσεις μεταξύ των θεσμοϊκών οργάνων στο μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουμε. Με κάθε σεβασμό και νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ποιε είναι οι αρμοδιότητες, πιστεύω ότι στο μέλλον θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι στενότερες δυνατές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό και στον τομέα της αεροπορίας με αμοιβαία ωφέλη Πρέπει λοιπόν στο μέλλον να υπάρξει συμφωνία στον τομέα τη αεροπορία, το βάζω σε εισαγωγικά γιατί δεν ξέρω αν θα είναι ξεχωριστή συμφωνία ή αν θα είναι ενταγμένη στη συνολική συμφωνία που ενδεχομένω είναι αυτή, αλλά πάντως θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελή για όλε τι πλευρέ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σχόλια που ήθελα να κάνω. Θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε αυτά τα θέματα, ιδίω βεβαίω των σκιωδών που είμαι βέβαιο ότι τα γνωρίζουν, αλλά Νομίζω ότι ε, αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τώρα αυτή τη στιγμή είναι να μάθουμε ποια είναι η θέση τη Κομισιόν, να, να πάρουμε αυτές τις διευκρινήσει που ανέφερα και να εξασφαλίσουμε ότι μαζί με το Συμβούλιο θα ε, υπάρχει στο μέλλον μια αμοιβαία εποφελής συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριε Τέλητσκα, κύριε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 να σας πω καταρχάς ότι το Brexit είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από το πώς θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και τα δύο μέλη οφείλουν να προετοιμαστούν σε, για ένα σενάριο σκληρού Brexit. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για μια έξοδο άνευ συμφωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και να ε, μπορέσουν να εγγυηθούν ε, μια συνέχεια ε, και μια ασφάλεια για την ε, ευρωπαϊκή αεροπλοεία, ούτως ώστε οι πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζουν να γίνονται με τα πιστοποιητικά που εκδίδει η ΕΑΖΑ και μετά από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να βρεθεί η λύση για συνέχεια. Είναι απαραίτητο οι φορείς να έχουν τον χρόνο που χρειάζονται στη διάθεσή τους για να μπορούν να χορηγούν τα πιστοποιητικά που ε, εκδίδονται με βάση το άρθρο 68 ε, του κανονισμού 2008-1039. Εγώ θα πρότεινα να εγκριθεί η πρόταση της Κομισιόν χωρίς τροπολογίες. Η δική μας ε, πρόταση είναι να τροποποιηθεί ε, η περίοδος, ε, η χρονική περίοδος για κάτι τέτοιο και είμαστε υπέρ οποιασδήποτε τροπολογίας παρατείνει αυτήν την μεταβατική περίοδο. Ε, ε, έγινε λόγος και για διαβούλευση του κοινού. Όμως δεδομένης ε, της, μάλλον του χρονικού περιορισμού πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Άρα λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις δυσκολίες, βασίζομαι στην καλή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές και αναμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελμόντε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αντίστοιχα πράγματα έχω να πω και για τις εμπορευματικέ μεταφορές. Είμαστε σε επιτυχημένη διαδικασία διότι πρέπει γρήγορα να εγκριθεί αυτό το, η μελέτη. Όλοι μας θέλουμε μελέτη αντικτύπου, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν για αυτή την πρόταση που εγγυάται τις βασικές ε, συνδέσεις για τις εμπορευματικέ μεταφορές και για την πρόσβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίω, θα ήταν καλύτερο να έχουμε καταφέρει νωρίτερα και να μην τοποθετηθεί αυτή η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο εν γέννη υπό τόσο μεγάλη πίεση. Πάντως, λήψη ε, συμφωνίας ε, πόσεση, οι υπηρεσίε μεταφορών εμπορευμάτων ε, ε, θα πρέπει να διέπονται από το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό δυστυχώς θα σήμαινε απώλεια γυρότητας των ε, κοινωνικών αδειών που χορηγούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο στους μεταφορείς των οδικών μεταφορών και κατά συνέπεια δεν θα υπάρχει πρόσβαση στην κοινή αγορά της και το ίδιο θα ισχύει και για τους μεταφορείς της Ένωσης προς τη Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν χρειάζεται να βρεθούν κάποια προσωρινά μέτρα που θα διέπουν τις εμπορευματικές μεταφορές ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφύγουμε έτσι από επιπτώσεις για τις Σύνδεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν ε, το βασικό είναι αυτό, ότι δηλαδή τα δικαιώματα που ε, δίνονται στους ε, μεταφορείς του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι αντίστοιχα με αυτά που δίνονται στους Ευρωπαίους μεταφορείς και αυτά που χορηγεί ε, το Ηνωμένο Βασίλειο στους Ευρωπαίους οδηγούς να είναι αντίστοιχα, ε, συγγνώμη, μεταφορείς να είναι αντίστοιχα. Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία. Στο άρθρο 4 βλέπουμε τι ισχύει τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 5 αφορά την αντιστοιχεία δικαιωμάτων με τη δυνατότητα η Κομισιόν να υιοθετεί κατ' εξοδότηση Και έχουμε και το άρθρο 6 ε, που προβλέπει παρακολούθηση από πλευρά τη Κομισιόν ώστε να υπάρχει εγγύηση πώς στηρούνται τα μέτρα αυτά θέμη του ανταγωνισμού και όλο το περιεχόμενο που μπορεί να έχουν αυτές οι κατεξοδότηση πράξεις με τη δυνατότητα φυσικά συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και δυνατότητα ελέγχου. Να ρωτήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει να, όταν λέει ή να υιοθετήσει σκόπιμα μέτρα, κατάλληλα μέτρα. Αυτή η διατύπωση είναι αόριστη και περιλαμβάνεται στο άρθρο 5, 5 όχι, συγγνώμη, παράγραφος 6, παρά, ε, άρθρο 6, παράγραφο 2 σε. <coughs> Με συγχωρείτε. Είναι ε, λέει εκεί την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων ε, που είναι κάπως αόριστο, ε, υπερβολικά αόριστο μάλλον και πρέπει να αποσαφενιστεί αυτή η διατύπωση. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και συνεδρίαση των σκιωδών και φυσικά και είμαι έτοιμη να συζητήσω και να δεχτώ προτάσεις από τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια για την παρουσίαση των ε, ευχαριστώ όλους τους εισηγητές για τις εισηγήσεις τους και θα δώσω το λόγο ε, ένα λεπτό έκαστος ε, για τις εκθέσεις ε, όλων, ε, για την έκθεση του κ. Τέλεσκα, ο κ. Δεγκράντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγος ο χρόνος, είναι απλοποιημένη διαδικασία, αλλά θα πρέπει να δώσουμε όλες μας τις ιδέες. Αλλά πρέπει ωστόσο να μπορέσουμε να το συζητήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για τη διαδικασία και όσο μπορώ πιο σύντομα θα κάνω πέντε παρατηρήσεις κάθετος ανησυχίες. Πρώτον, η ημερομηνία αναφορά. Ε, τόσο η αεροπλοεία όσο και ο τουρισμός και οι δύο τομείς συμφωνούν στο εξής, ότι δηλαδή το 2018 ως αναφορά ως έτος αναφοράς είναι πολύ αμφισβητήσιμο. Έπειτα, ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν ε, κατάλληλοι κωδικοί ε, όσον αφορά τις μεταφορικές ε, εταιρείες επιβατών. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών. Κανονισμός για τα αεροσκάφη διμερείς συμφωνίες που απαγορεύει η Κομισιόν με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, η Κομισιόν ορίζει τα δικαιώματα κυκλοφορίας των αεροσκαφών και μπαίνει στα εθνικά χωράφια. Στο κανονισμό 1008 του 2008 θέλω να, ζητήσω, να ρωτήσω το εξής να συμπεριληφθεί αυτό το σημείο σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, η ισχύ των αδειών εξαγωγών είναι το βασικό στοιχείο για να μην επηρεαστούν οι ευρωπαϊκές εμπορευματικές, ε, ε αεροπορικές μεταφορές, γιατί έτσι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα όσον αφορά τις πτήσεις, ακυρώσεις κτλ. Υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση για τον κανονισμό 1008-2008. Τι νόημα έχει λοιπόν να επιβάλλουμε κριτήρια τα οποία μπορεί στη συνέχεια πάλι να αλλάξουν. Άρα λοιπόν προτείνω το εξή. Παράταση της ισχύω των, ε, των ε, εγκεκριμένων αδειών για ακόμα ένα χρόνο μέχρι ότου να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ε, θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε Δεγκράν. Το ξέρω πως ε, είναι πιεστικό αλλά τι να κάνουμε. Κυρία Φώστερ, έχετε εσείς το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Και εγώ νομίζω πως θα ε, ξεπεράσω το ένα λεπτό, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα αρκετά που είπαν ε, οι ομιλητές και ο προηγούμενος ομιλητής. Δεν έχει ληφθεί υπόψη, νομίζω, πως υπάρχει 6% αύξηση της και κυκλοφορίας ε, για το 2018, για το οποίο είχε προτιμιστεί εκ των προτέρων Ευρωκοντρόλ, οι αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες ελέγχου, ελέγχου κτλ. Α, τώρα, αν μόνο αν κάποιο κάτσει και παίρνει τηλέφωνο έναν έναν όλους του πελάτε να του πει ότι ακυρώνονται οι διακοπέ του, μπορεί κάτι να γίνει. Έχουμε την ΙΑΤΕ, τη ΤΟΥΗ που είναι ένα πολύ μεγάλος, μια πολύ μεγάλη εταιρεία και ανησυχεί φοβερά, διότι πέντε από τις χώρες, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, μπορεί να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν με βάση τους κανόνες που φτιάχνονται τώρα. Εγώ θα ήμουν υπέρ του να υπάρξει συμφωνία, να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση, είτε είναι προσωρινή είτε όχι. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι έχουν, προβλέπονται 5 εκατομμύρια έξτρα θέσει στο σύστημα αυτό το καλοκαίρι και ένα τέταρτο αυτών αφορά το ε, τουρισμό ανάμεσα Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Για πείτε τα αυτά στον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμό της Ισπανίας. Τέλος, απογοητευτικό επίσης είναι ότι και οι Αμερικανοί έχουν ε, εδώ δίκιο. Δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε σε έναν ε, νέο ε, ανοιχτό ουρανό οι Αμερικανοί λοιπόν δυσαρεστούνται πολύ με τα όσα βλέπουν εδώ, γιατί ξέρουν ότι αυτά που προτείνεται κατα... παραβιάζει τη συμφωνία ανοιχτών ε, ουρανών ανάμεσα στι ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να προτείνω λοιπόν Κομισιόν να πάτε πάλι στα γραφεία σας και να τα ξανασκεφτείτε και να προσπαθήσετε να λύσετε αυτά τα θέματα, γιατί θέλουμε να μείνουν απλά τα πράγματα δεν θέλουμε να, να αποφύγουμε τη συμφωνία, να τα αποφύγουμε όλα αυτά. Ας βάλουμε λοιπόν, ας κάνουμε πρακτικές προτάσεις, γιατί πραγματικά αυτό εδώ είναι πολύ απογοητευτικά. Εδώ και χρόνια έχω να δω τόσο πολύ χάλια πρόταση. Κοιτάξτε, άμα όλοι μιλάτε για δύο λεπτά θα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις τρεις, άρα δεν γίνεται. Μπείτε λοιπόν στην ουσία. Euh, Νταλούνται, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα ε, μακρηγορήσω. Είδα τις ε, προτάσεις και γενικά ε, συμφωνώ με τη θέση της Κομισιόν ακόμη και αν ε, θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να μας είχαν δώσει τη δυνατότητα να το εξετάσουμε περισσότερο χρόνο, θα μπορούσαμε να μα το έχουν δώσει πιο νωρί την πρότασή τη γιατί θα ήμασταν σε καλύτερη θέση. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχω κάτι να ε, πω για την, ε, για την ουσία της πρότασή του. Σας ευχαριστώ και περνάμε τώρα στην έκθεση Ζωτόσκη και δίνω το λόγο στον κύριο Γίγκολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στηρίζω το, γεγοντό, το γεγονός ότι η Κομισιόν μετά την ε, απόρριψη της συμφωνίας από το Βρετανικό Κοινοβούλιο επανεξετάζει τις προτάσεις αυτές. Εδώ για την ασφάλεια της αεροπορίας νομίζω ότι το θέμα δεν είναι ακανθόδες ε, ούτε θα δημιουργήσει προβλήματα αν και δεν είχα την ευκαιρία και εγώ να συζητήσω με τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους φορείς γι' αυτό και θέλω να είμαι προσεκτικός και σύντομος. Η διατήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας, ακόμη και σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης της ε, Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητος όρος. Να πω επίσης ότι ε, μια ε, δυσαρμονία ή μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τις υποχρεωτικές απαιτήσει ασφαλείας, ασφαλείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα και στους Ευρωπαίους αεροναυπηγούς. Βεβαίως το θέμα αυτό σχετίζεται με την ασφάλεια αλλά σχετίζεται και με την οικονομία και με τις θέσεις εργασίας. Γι' αυτό και ε, θεωρώ ότι η πρόταση κομμεσιών ευτυχώς στη βάση, του και στο πνεύμα, στο, στη βάση της και στο πνεύμα της ε, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι απαραίτητο η Βρετανία και μετά το Brexit να διατηρήσει την ισχύ και την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας για να εξασφαλίζεται και η συμμόρφωση και η συμβατότητα όλων των συστημάτων και στο μέλλον και γι' αυτό ε, υποστηρίζω ε, ε, την πρόταση της Κομισιόν η Βρετανία να θεωρείται τρίτη χώρα υπό την ευθύνη της ΕΑΣΑ. Ο κύριος Τέλιτσκα θα την καταστήσει τον κύριο Βαντενμπουργκ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, ο συνάδελφος δεν μπορούσε να είναι εδώ, αλλά θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό να σας πω αυτά που θέλει να σας πω. Ο κύριος Βαν Μίλτεν λέει ότι είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο χαιρετίζει την πρόταση για ομαλή αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση να σημειωθεί ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι όροι της αποχώρησης της Βρετανίας ε, να εξασφαλίζουν την συνέχιση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συντήρηση, την επισκευή και την κατασκευή αεροσκαφών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να, εξασφαλιστεί, ε, να εξασφαλιστούν τα αμοιβαία συμφέροντα Βρετανίας και Ένωσης. Πάντως θα πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλό και ομοιογενές επίπεδο προδιαγραφών ασφαλείας, ακόμη και αν η Βρετανία γίνει τρίτη χώρα θα πρέπει να οδηγηθούμε σε όχι λιγότερες αυστηρές, ε, αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας. Ευχαριστούμε κύριε Τέλιτσκα. Τέιλορ. Κύριε Τέιλορ. Και για την ΚΟΕ δεν είναι εδώ η πρόσωπος, οπότε περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ντεμόντε με τους κοιόδες της. Κυρία Κλούν. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε ότι με το θέμα αυτό ασχολούμαστε εδώ και καιρό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία εκτό ανάγκη, διότι ε, πρέπει να υπάρχει μια λύση σε περίπτωση που χρειαστεί. Νομίζω οι διμερείς μεταφορές είναι μια λύση και σχετικές συμφωνίες και αυτό να δημιουργήσει ε, την δυνατότητα να καλυφθεί το χάζα μεταξύ της Βόρειας Ισλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και Απλώς θα πρέπει να βελτιώσουμε κάπως το σχετικό ορισμό. Ας πούμε, πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η διέλευση από την Ευρώπη προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Καλέ και ποιες θα είναι οι ρομεταφορές ποιες θα είναι οι που θα περνούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Πρέπει να το πούμε ε, για να δουν τι θα κάνουν και οι αερομεταφορεί και του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ευρώπη και θα πρέπει και για το καμποτάζ να προβλέψουμε σαφεί κανόνε για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά είναι συμβατά με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλούν. Κύριε Σλοτόφσκι, έχετε το λόγο. Για την κυρία Ντεμόντα. Ευχαριστώ. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές το πλέον σημαντικό είναι η δυνατότητα όλες οι υπηρεσίες μεταφορών να μπορούν να προσφέρονται με τον ίδιο τρόπο ε, και μετά τον Brexit. Καμποτάζ, ε, διέλευση χωρίς εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά. Διότι ιδάλλως ε, θα πληγούν εταιρείε και δεν θέλουμε, ιδίως για αυτές που παρέχουν υπηρεσίε στον Ηνωμένο Βασίλειο. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι γραμμές λεωφορείων. Έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις για τα λεωφορεία και τα πούλμαν λειτουργούν και πέραν του Brexit, αλλά εάν υπάρξει αποχώρηση, ε, θα υπάρξει και αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από αυτέ τι συμφωνίε. Δηλαδή, μεταφορά επιβατών δεν θα είναι πλέον εφικτή, διότι δεν θα υπάρχει νομική βάση. Αυτό πραγματικά θα πλήξει τι εταιρείε που προσφέρουν τέτοιε εταιρείε. Ελπίζω λοιπόν ότι στην απογευματινή μα συνεδρία θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, ευχαριστώ την Επιτροπή γιατί είναι περίπλοκο ο ρόλο τη. Όντω, κανένα μα δεν ξέρει τι θα συμβεί και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε προτάσεις ενώ, ενώπιον ενός αβέβαιου ε, μέλλοντος όπως βλέπουμε τα εξάλλου τις τελευταίες εβδομάδες και μέρες. Πιστεύω πως φέρουμε την ευθύνη να προχωρήσουμε για να δώσουμε την ασφάλεια στον τομέα αυτό, να προσφέρουμε ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια τα οποία να ζημιώσουν όχι μόνο τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό το τομέα αλλά και, και, για να μπορούμε να πούμε πως οι μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει όντως να προβλέψουν τα πράγματα γιατί εφόσον έχουν τακτικές ε, μεταφορές με το Ηνωμένο Βασίλειο να έχουν άδειε ώστε να μπορούν να ε, συνεχίσουν να εργάζονται. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υιοθετήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για να αποφύγουμε όλες αυτές τις επιπλοκές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βελπάο. Κύριε Τέιλορ, ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος Ό,τι και αν πιστεύει κανείς για την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για απόσυρση που πιστεύω πως είναι απίστευτα ανόητη και καταστροφική, ήρθε αυτό εμπαρόδο, Νομίζω πως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ισότιμο πεδίο τόσο για τους Ευρωπαίους όσο και για τους Βρετανούς μεταφορείς. Ο αντίκτυπος ε, για τις ε, οδικές επαγγελματικές μεταφορές ε, προκαλεί ανησυχίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την επιθεώρηση τροφίμων και ε, ζωοτροφών ε, στα σύνορα. Θα ήθελα να μπορέσουμε να μελετήσουμε την πρόταση καλύτερα και να σκεφτούμε την υποβολή πιθανών ε, τροπολογιών. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Είχαμε τους σκιώδεις συγητές, τους ακούσαμε για τα σημεία κλειδιά και τώρα θα ακούσουμε την Κομισιόν, κύριος Κορνέλης και η κυρία Βένερ που θα μιλήσουν για το σύνολο των σημείων αυτών. Έχετε το λόγο, παρακαλώ λίγο σύντομα, γιατί καθυστερήσαμε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω για τα δύο κείμενα περί αεροπλοίας και όπως είπατε, η συνάδελφος, η κυρία Βέρνερ, θα μιλήσει για τις οδικές. Να θυμίσω ότι ε, ο μόνος στόχος της πρότασης για τα έκδοτα μέτρα είναι για να αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες που θα προκληθούν στην Ευρώπη των 27 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Δεν είναι ένα σενάριο που θα θέλαμε να ε, γίνει πραγματικότητα, όμως μπορεί να συμβεί λόγω των, των αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού και δεν ελέγχουμε. Ε, η μόνη δυνατότητα είναι να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε το αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Είναι σαφές ότι τα μέτρα και το σύστημα που προτείνονται ως συνέπεια λόγω των έκτακτων μέτρων δεν μπορούν καθόλου να επιτρέψουν την αυτόματη συνέχιση της, της κατάστασης που επικρατεί σήμερα λόγω της ισχύω της ενιαίας αγοράς και του συστήματός της. Τα δικαιώματα, η πρόσβαση θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντική συμφωνίας. Δεν μπορούν να ισχύουν αυτομάτως το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα. Αυτά θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση στο μέλλον. Το να προσαρμοστούμε σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία είναι καθήκον κάθε πολίτη και κάθε επιχείρηση. Σε πολλαπλές περιπτώσεις έχουμε ενημερώσει επιχειρήσεις και πολίτες για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που ε, έχουμε τέτοιο Brexit. Τους έχουμε πει τι προσαρμογές μπορεί να χρειαστούν. Έχουμε εκδώσει πολλά ενημερωτικά φυλάδια, έχουμε διοργανώσει ενημερωτικέ εκστρατείες και σε επίπεδο ΕΑΖΑ και όχι και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι να περιμένει. Αυτή είναι η πρώτη αρμοδιότητα και καθήκον που έχουν όλοι, να προετοιμαστούν. Ε, τα μέτρα, τα έκτακτα μέτρα, σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τι περιπτώσει όπου οι ιδιώτε δεν μπορούν να έχουν προετοιμαστεί για τον οποιονδήποτε λόγο εγκαίρω. Οπότε, για το κείμενο που αφορά την ασφάλεια, ίσως πρώτα. Εν είδη παραδείγματο για, την, ε, για τα επίπεδα προετοιμασία, έχουμε πει στου πιλότου στην Ευρώπη, στου πιλότου που έχουν ε, βρετανικέ άδειε άσκηση επαγγέλματο, ότι θα πρέπει να τι ε, αλλάξουν και να πάνε σε ένα ευρωπαϊκό κράτο. Να σα βεβαιώσω ότι μηχανικοί πιλότοι και πλήρωμα αεροσκαφών, κατά εκατοντάδε το έχουν κάνει αυτό. Τα έκτακτα μέτρα αφορούν πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, όπως κάποια τμήματα αεροσκαφών να έχουν χαλάσει μετά το Brexit και να μην μπορούν να αντικατασταθούν. Ε, είναι ένα παράδειγμα. Ε, Νομίζουμε ότι έχουμε καλύψει όλες τις δυνατές περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν ως προς την προετοιμασία ή τα έκτακτα μέτρα, διότι δεν είχαμε περαιτέρω αιτήματα ούτε στο Συμβούλιο ούτε στις συζητήσεις μας για να προσθέσουμε κάτι ακόμα και να σας πω ότι στις συζητήσεις του Συμβουλίου κάποιο ίσονο σημασίες διορθώσεις και αποσαφηνήσεις χρειάστηκαν αλλά δεν άλλαξε το πνεύμα της προσέγγισής μας σε καμία περίπτωση. Και Περαιτέρω συζήτηση γίνεται σήμερα στο Συμβούλιο την ώρα που μιλάμε. Πρότασή μας θα ήταν τις διορθώσεις και τις αποσαφηνίσεις που θα θέλετε από την πλευρά του Κοινοβουλίου να τι κάνετε κατά τρόπο ώστε να γίνει ευκολότερη και ομαλότερη όλη η διαδικασία έγκριση τη πρόταση Τώρα για την πρόσβαση στην αγορά και το σχετικό θέμα. Σημειώνω τις παρατηρήσεις του κυρίου Τέλιτσκα και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ελευθερίες από τις τέσσερις που αναφέρονται εδώ για τις πτήσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή περαιτέρω απελευθέρωση στο σύστημα θα είναι αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων ούτως ή άλλως. Για το θέμα της ε, ιδιοκτησία και τη ανάληψη ευθύνη που τέθεσε πάλι ο κύριο Τέλιτσκα, θεωρούμε ότι είναι ένα θέμα όπου οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν. Το καλοκαίρι του 2017 συζητήθηκε αυτό σε δημόσιες διαβουλεύσεις και σας διαβεβαιώ ότι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία τους και είναι πανέτοιμες μπορούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες ελέγχου. Γι' αυτό δεν βλέπουμε να χρειάζονται ειδικέ διευθετήσει. για το θέμα του όγκου της κυκλοφορίας η συλλογιστική μας, όπως ρώτησε και ο κ. Στέλιτσκα, ήταν ότι από τη στιγμή που μιλάμε για έκτακτα μέτρα, ο στόχος θα πρέπει να είναι να έχουμε βασική διασύνδεση για το προς των επιχειρήσεων και των επιβατών, των πολιτών, για να μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ συγκεκριμένων ε, γεωγραφικών σημείων. Ο όγκος λοιπόν των μεταφορών ε, του 2018 θα πρέπει να παραμείνει ίδιος και στο μέλλον. Ακόμη και αν δεν υπάρξει συμφωνία. No deal Brexit. Αυτό ήταν το σημείο εφετερία μας. Ο κύριο Τελίτσκα ανέφερε το θέμα της ημερομηνία. Υπάρχει ημερομηνία στην Αντολή για τα μέτρα πρόσβαση στην αγορά και τη σχετική πρόταση και ακολουθεί τις εποχές της ε, ε, ΙΑΤΑ όπως ονομάζονται. Νέα μήνες είναι η τωρινή μας πρόταση ώστε να έχουν τη δυνατότητα όσοι κρατούν ε, άδειες και πιστοποιητικά του Ηνωμένου Βασιλείου να πάνε στην ΕΑΖΑ και να μπορέσουν να τα πιστοποιήσουν ως πιστοποιητικά και άδειες τρίτης χώρας. Τώρα έγινε αναφορά στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα, Πρόθεσή μας είναι να σεβαστούμε πλήρως τις υποχρεώσεις μας βάσει της συμφωνίας αυτής και οποιασδήποτε άλλη εξωτερική συμφωνίας ε, σε κάθε περίπτωση και δεν έχουμε ενδείξεις ότι οι ομόλογοι μας από τις ΗΠΑ έχουν εδώ διαφορετική άποψη. Ε, θα πάψω εδώ, Πρόεδρε, και θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις Απλώς να επισημάνω ότι θα πρέπει να ε, ανασκουμποθούμε, διότι είναι δικό μας φάρμα που ήρθαμε τόσο αργά να σας προβάλλουμε την πρόταση αυτή, αλλά όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε, τόσο πιο γρήγορα και τα κρατικά συστήματα των κατωμελών θα μπορέσουν να δώσουν τις σχετικές άδειες και ε, πιστοποιητικά στι αεροπορικέ εταιρείε, γιατί αυτά είναι αναγκαία. Ε, Παθιόμαστε λοιπόν στην ε, ενεργή και επικοδομητική σα συνεργασία ε, για να περάσει το θέμα κατεπηγόντω. Και είμαστε στη δίδασή σα για να σα βοηθήσουμε. Και σε εσά και στου εισηγητέ, εφόσον χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βεντέρ, πολύ γρήγορα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο Φίλιπ ως γενικά σχόλια για τα επόγοντα μέτρα και για τη διαδικασία. Πρέπει να ακολουθήσουμε την επιτυχημένη διαδικασία. Στην οδικέ ε, μεταφορές είδαμε ποια θα ήταν η εναλλακτική και ποια θα ήταν η εναλλακτική όσον αφορά τις, τα μερίδια, τα, τις και το ECM Forum ε, αποφασίσαμε ότι δεν θα ήταν ε, επαρκές, γι' αυτό και ε, προτείναμε να συσταθεί ένα προσωρινό φόρουμ, μέσω του οποίου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δίνονται προσωρινά δικαιώματα ώστε να μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει μια ελάχιστη εναέρια κυκλοφορία και να υπάρχει μια συνδεσιμότητα αλλά για περιορισμένο πεδίο και ε, χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παράσχει στην ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα στις εμπορευματικές εταιρείες να μεταφέρουν εμπορεύματα υπό όρους όμως ε, που θα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να παράσχει αντίστοιχα ε, δικαιώματα στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές κοινωνικές, εργασιακές και να εξασφαλίζεται ο δίκαιος και θεμητός ανταγωνισμός. Θέλω να το εξηγήσω. Επειδή θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία επικράτεια, ένα τέτοιο μέτρο θα επέτρεπε το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ και των κρατών μελών και όλων των κρατών μελών ως σύνολο με, το, με την Βρετανία και αντιστρόφως. Αυτό δηλαδή δεν έχει καμία επίπτωση στην εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα, όσον αφορά ε, τα ερωτήματα ε, De Υπάρχει διάταξη η οποία επιτρέπει στην Κομισιόν να παρακολουθεί τα δικαιώματα και φυσικά ζητεί ε, από την Κομισιόν να παρακολουθεί αυτά τα δικαιώματα και να εξασφαλίζει ότι ε, υπάρχει ίσως όρος, ε, ίση όρη ανταγωνισμού και θεμητό ανταγωνισμό. Και η Κομισιόν μπορεί να λάβει μέτρα σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και εδώ θέλω να σας πω ότι συγκεκριμένα έχουμε προβλέψει θα προχωρούσαμε σε αναστολή αυτών, των διατάξεων μόνο εφόσον ε, διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα ως προς την εφαρμογή αυτών των ε, κανόνων. Θα μπορούσαν όμως να οριστούν και ε, κάποια όρια όσον αφορά τη χορτικότητα ή τον αριθμό των ταξιδιών ή θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποιες επιχειρησιακοί περιορισμοί τους οποίους έχουμε προβλέψει. προβλέψει. Να απαντήσω και στην κυρία ε, Κλούν για τη διέλευση στην ενωσιακή επικράτεια, για μας είναι σαφές ότι εφόσον ε, ε, ε, ότι για μας η, η Ιρλανδία καλύπτεται. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούν εμπορεύματα να μεταφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Βρετανίας και πάλι πίσω σε επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιρλανδία. Για το καμποτάζ. Για μα αυτό δεν είναι ζήτημα δημόσια τάξη, γι' αυτό και δεν καλύπτεται από αυτή την πρόταση. Είναι προφανέ ότι ε, αυτό δεν είναι ισοδύναμο με την ενιαία αγορά, ούτε μπορεί να εξασφαλίσει από μόνο του την συνέχεια τη ενιαία αγορά. Αυτό θα γίνει μόνο αν ε, καταρτιστεί και συμφωνηθεί μια νέα σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και ε, ρωτήσατε και για την μεταφορά κωδικών επιβατών. Εδώ υπάρχει ε, μία ε, πρόταση ενδιάμεσης συμφωνίας, ώστε ε, τη συμφωνία μάλλον Interbus, στην οποία μπορεί να προσχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, άπαξ και καταστεί τρίτη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω ότι στις διαδικασίες έχουμε απόψε τους σκιώδεις ε, εάν υπάρξουν τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν στο όνομα της Επιτροπής και άρα στον εισηγητή πριν τις 24 Φεβρουαρίου. 24 Ιανουαρίου, συγγνώμη. Άρα δηλαδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Στη συνέχεια έχουμε 24 Ιανουαρίου ξεκινά μια, ένα δεκαήμερο που εκεί μπορεί κανείς να καταθέσει ενστάσεις. εκτός αν υπάρξουν αντιρρήσεις. Οπότε το σύνολο των συμφωνιών θα ψηφιστούν στις 4 Φεβρουαρίου, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, ο στόχος είναι 29 Μαρτίου του 19 όπου οι Άγγλοι δυστυχώς θα μας αφήσουν. Αλλά πριν θα πρέπει να έχουμε αυτές τις συμφωνίες στην επίσημη εφημερίδα. Οπότε όλοι έχουμε βάλει ε, τε, μπρος, έχουμε ανασκουμποθεί. Αυτά λοιπόν για το Brexit. Και τώρα θα ψηφίσουμε... Si nous avons atteint le quorum. Εδώ αν έχουμε απαρτία. Allez, euh, λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν με την απαλλαγή. Bon. Allez, on commence par le rapport de Monsieur Franck Prouveau sur... Allez, le rapport de Monsieur Prouveau sur les décharges 2017. Έκθεση του κυρίου Προύστου για την απαλλαγή. Υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Υπέρ, τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Σοσιαλιστές έχετε έναν παραπανίσιο. Πέρα στην ψηφοφορία. Plus 35, Contre 6. Bravo, monsieur Franck Prouveau, vous lui direz. Ε, μπράβο σας, εγκρίνεται η έκθεση κύριε ε, Προύστ. Πάμε στην έκθεση στη Λεοντίνη. Shift to Rail. Τροπολογία 1. Περ κατά. Είμαστε στο Shift to Rail, παιδιά. Τι θέλετε να αρχίσουμε από την έμσα. Άντε, ας αρχίσουμε από την έμψα Allez, on commence par l'Agence européenne du maritime. Ε, Ευρωπαϊκός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Τροπολογία 1, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα γιατί είναι ακριβώς τι σημαίνει τι ισχύει οπότε θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά άρχεται για το 6 για την τροπολογία 6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 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Je ferme le vote.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 Ψηφίζουμε για την 6 ηλεκτρονικά. Τέλος. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, ναι Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου για την ΕΡΑ. Τέλος της ψηφοφορίας. Και το κείμενο εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα πάμε στο Shift to Rail, το Cesar. Τροπολογία 1. Α, ναι, είτε είναι το ένα είτε είναι το άλλο, θα εγκριθεί, θα το ψηφίσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Σέζαρ. Ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το κείμενο. Τέλος. Και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συνεχίζουμε με το Shift to Rail. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε τέλος και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα κείμενα που εγκρίθηκαν για τις απαλλαγές για τους διάφορους οργανισμούς και τώρα περνάμε στην πρόταση απόφασης Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που τοποποιεί την, την ε, Οδηγία 96 του Συμβουλίου σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων για το μέγιστο μήκο στην περίπτωση θαλάμων οδήγηση που παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα ω προ την αεροδυναμική απόδοση, mm. τη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τι επιδόσει ασφάλεια. Εγώ είμαι η συγχύτρια τροπολογία 1 υπέρ. Την έχετε? Είμαστε στην έκθεση Καρίμα Ντελή. Το βρήκατε. Allez, on y va. 1 qui est pour. Qui est Υπέρ κατά αποχές. <laughs> Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του κειμένου. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Μπράβο σας κυρία Ντελή. Allez, on va voter le mandat de négociation aussi. J'ouvre le vote sur le mandat de négociation. Τώρα, διαπραγματευτική εντολή. Ψηφίζουμε. Ouvert le vote. Τέλος. Και η διαπραγματευτική εντολή λοιπόν εγκρίνεται με, μεγάλη πλειοψηφία. Et nous continuons sur le rapport de M. Zille sur l'accès au marché. Έκθεση Ζήλε. Κοινοί κανόνε πρόσβαση στα διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία. Allez, on Πάμε. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 37. Πέρας. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο, υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές Ακόμα και αν έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Να έρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Τι ψηφοφορία. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία για την απόρριψη. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, Εποχές. εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 130. Υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση. 130 πέρας. Α, έχετε δίκιο. Αγκρίθηκε. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. 171 και 172 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Επαλήθευσης. Άρχεται η ψηφοφορία για τις δύο τροπολογίες, και 171-172. Ε, πέρας. Απορρίπτονται. Τρεις ταυτόσημες, 173-175 υπέρ. Κατά, εποχές, απορρίπτονται. Ταυτόσημες, 176-177 υπέρ. Κατά, Αποχές. απορρίπτονται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτεται. Ταυτόσημες, 179-180 απορρίπτεται. 10, συμβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη συμβαστική 11. 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο ταυτόσημες. 2.31, ε, 2.32, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ε, συμβαστική 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απευθείας συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 329 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές. να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με διαφορά. Πηγαίνουμε απευθεία στη συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 371 ταυτόσημη με την 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν σαφές. 36. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. Εγκρίνεται. 18, συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές. Πάλι δεν είναι σαφές να ξαναψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. 18, παρακαλώ. Κάποιος είναι περάριθμος. Πέρας, η συμβαστική 18 εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 383. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 390 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 391 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 395 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 394. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 396. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 397. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 397 επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Σε Ξεκάθαρα. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46, τροπολογία 46, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται να επαληθεύσουμε για την 58. Πέρας. Γκρίνεται. Έχετε δίκιο, κύριε Κόχ. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. απολύτω. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, εποχές δεν σαφές ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 89 παρακαλώ πέρας εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Ζήλε. Η έκθεση εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Μπράβο σας κύριε Ρόμπερτ Ζήλε. Allez, il y a encore un vote, Δεν τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Για καθίστε κάτω, συγκεντρωθείτε. Μένει μια ψηφοφορία. Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη ψωνόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Συνθήκη για την Ίδρυση Κοινότητα Μεταφορών. Υπέρ. Α, ηλεκτρονικά να με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Και εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Μπράβο συνάδελφοι, ευχαριστώ. Και θα περιμένουμε τώρα την Ρουμάνα Υπουργό για να έχουμε διάλογο με την Υπουργό που θα έρθει. Οπότε θα διακόψουμε για 10 λεπτά. Έχουμε 10 λεπτά διάλειμμα. Je vous donne rendez-vous. Ραντεβού ευθύς από... La commission n'est pas encore là. Nous nous, nous, nous retrouvons à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

Συνάδελφοί μου, να ξεκινήσουμε. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Είναι μεγάλη τιμή να σας υποδεχόμαστε εδώ, κυρία Υπουργέ, των μεταφορών, κυρία Ροβάνα Πλούμπ, ε, θα μας ε, αναπτύξετε τις μεγάλες προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Ξέρετε, από την 1η Ιανουαρίου η Ρουμανία ανέλαβε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, και με πολλές φιλοδοξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς έχουμε μάθει ότι για τις μεγάλες σας προτεραιότητες υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες. Η κινητικότητα και η φόρος βιωσιμότητα. Εδώ βλέπουμε ότι θα υπάρχουν τότε συνέπειε για τους Ευρωπαίου πολίτε και για την κοινή αγορά. Και θέλουμε να μειωθούν οι αποκλήσει και οι ενισότητες μεταξύ των διαφορών περιοχών, να γίνουν μαζικέ επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ότι όλα αυτά ε, μας φέρνουν στην θέση κοινών στόχων για τα κοινά μας συμφέροντα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ της Προεδρίας και της Επιτροπής μας. Σας εύχομαι κάθε τύχη για το εξάμεινο τη Ρουμανικής Προεδρίας. Θα σα δώσω 15 λεπτά για να μας παρουσιάσετε τις μεγάλες σα προτεραιότητε. Και μετά θα έχουμε συζήτηση με τους συντονιστές και τα μέλη της ομάδας. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Mm. Ευχαριστώ κυρία Ντελή, ευχαριστώ πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους και θα ήθελα να σας πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον τομέα των μεταφορών. Έναν από τους πιο ε, σημαντικούς ε, κλάδους και τομείς και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Για να ξεκινήσω θα ήθελα να σας παρουσιάσω το πλαίσιο και τους γενικούς στόχους της Ρουμανικής Προεδρίας. Η Προεδρία μας ε, δίνει έμφαση στις ευρωπαϊκές αξίες και στην υποστήριξη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε αυτό το ε, ευρωπαϊκό εγχείρημα μέσω δημόσιων πολιτικών τις οποίες θα προωθήσουμε από κοινού. Η Προεδρία μας έχει θέσει στο επίκεντρό της τον πολίτη. Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών μας και να είμαστε πιο ρεαλιστές. Θέλουμε να έχουμε έναν δίκαιο διάλογο μαζί σας και με με εσά, ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είμαστε ένας ειλικρινή συνομιλητής και παράγοντας διευκόλυνση της συνένεσης. Η Προεδρία μα, όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, είναι φιλόδοξη και ρεαλιστική ταυτόχρονα. Φιλόδοξη διότι θέλουμε να προχωρήσουμε πολλά θέματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ξεκινώντας τριμερείς διαλόγους με και ρεαλιστές επειδή ενώπιόν μας έχουμε πολλές προκλήσεις όπως είναι το Brexit, οι ευρωεκλογέ και το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σύνθημα της Ρουμανικής Προεδρίας είναι «Συνοχή, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία». Και αυτή θα είναι η αρχή επί της οποίας θα βασίσουμε τις δράσεις μας σε όλους τους τομείς. Η πλατφόρμα της, προ... της Προεδρίας μας ε, συμπεριλαμβάνει τέσσερις πυλώνες. Την Ευρώπη της σύγκλησης, μια ασφαλέστερη Ευρώπη, μια Ευρώπη ως ισχυρός ε, παγκόσμιος παίκτη και μια Ευρώπη κοινών αξιών. Ο κλάδος των μεταφορών ε, ανήκει στον πρώτο πυλώνα, την Ευρώπη της σύγκλησης. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Οι πολιτικές στον τομέα των μεταφορών συμβάλλουν στην εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συνοχής και σύγκλησης για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης, της συνδεσιμότητας, της, ψηφια... της ψηφιοποίησης και της βιώσιμης ε, πολυτροπικότητας, στοιχεία που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα. Και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου ε, προς τις προηγούμενες προεδρίες για το έργο τους. Όλες οι προηγούμενες προεδρίες μαζί με εσά βεβαίω συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τη ενιαία αγορά καθώ και στην ανάπτυξη μια ολοκληρωμένη ανταγωνιστική πολυτροπικής και ε, ασφαλούς δικτύωσης μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις επιπτώσεις που έχουν οι μεταφορές στο περιβάλλον και θέλω να σας, ε, να σας διαβεβαιώσω ότι η Ρουμανική Προεδρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις, ε, στις νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν στον τομέα των μεταφορών που συζητιούνται φέτος, όπως είναι για παράδειγμα ε, το σενάριο μη ύπαρξη συμφωνίας για το, για το Brexit. Στο πλαίσιο αυτό ε, μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση του Brexit για, τις, ε, για την αυτιλία. Χθες το βράδυ καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, προωθούμε την διαπραγμάτευση ε, στα τρία πακέτα της κινητικότητας για να επιτύχουμε έναν δίκαιο συμβιβασμό όπου αυτό είναι δυνατόν, στον τομέα των χερσαίων, υδάτινων μεταφορών και των αντίστοιχων υποδομών. Και τώρα θα ήθελα να συνεχίσω στην ε, μητρική μου γλώσσα. Στον τομέα των ε, οδικών μεταφορών θα πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη το θεμητό ανταγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τι ανάγκες της αγοράς και χωρίς ε, περιττό διοικητικό φόρτο. Είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν οι κοινωνικές συνθήκες ε, των εργαζομένων, να βελτιωθεί το επίπεδο της ε, οδικής ασφάλειας ε, να καταστεί πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος αλλά και η τήρηση των ε, κανόνων να επιβληθεί όσον αφορά τον κοινωνικό πυλώνα το Συμβούλιο έχει επιτύχει τη γενική προσέγγιση παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση του Κοινοβουλίου και είμαστε διαθέσιμοι για συζήτηση Ταυτόχρονα ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μαζί σας για τα ε, νοικιαζόμενα αυτοκίνητα που είναι κομμάτι του πρώτου πακέτου για την κινητικότητα και το οποίο έχει συντάξει ήδη έκθεση το Κοινοβούλιο. Θα καταβάλουμε τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε το Συμβούλιο να μπορέσει να συζητήσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο για αυτό το θέμα και έτσι στη συνέχεια να μπει σε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σας. Σκοπός είναι λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Η ασφάλεια, οδική ασφάλεια. Πρόκειται για έναν ε, στόχο προτεραιότητας της Ένωσης. Ε, γι' αυτό και το θέμα της διαχείρισης των οδικών υποδομών είναι θέμα κλειδί για την Προεδρία της Ρουμανίας. Ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες διαφορές ανάμεσα στους συνομοθέτες όσον αφορά ας πούμε, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ή το σύστημα σήμανσης και ε, ε, το σύστημα σήμανσης θα ξεκινήσουμε από αύριο το διάλογο για να ε, μπορέσουμε γρήγορα να ξεπεράσουμε τις διαφορές ε, και για να πετύχουμε συμφωνία μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου. Τώρα, σε σχέση με την απόφαση για την ημερομηνία την προθεσμία μάλλον για την προσαρμογή των θαλάμων οδήγησης αεροδυναμικής ε, κατασκευής και αυτό το θέμα για μας αποτελεί προτεραιότητα γιατί πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εκ πρώτης όψης είναι πολύ απλή αλλά θα επιτρέψει την μείωση της κατανάλωσης ε, καυσίμου την μείωση των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα το, τη μείωση του κόστου των μεταφορών και ταυτόχρονα την, ε, θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Στο δεύτερο τμήμα της ε, θητείας μας θα θέλαμε να προχωρήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις όσον αφορά με την Ευρωβινιέτα και το δικαιώματα των επιβατών στις σιδηροδρομικές μεταφορές ώστε να υπάρξει πραγματική πρόοδο στο Συμβούλιο. Για τις ε, διατροπικές μεταφορές θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ώστε να πετύχουμε μαζί σας μια συμφωνία για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένε μεταφορές. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για τον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών και ελπίζουμε ότι ε, στον επόμενο τριμερί θα πάνε καλά τα πράγματα. Επίσης ε, θα θέλουμε να προσέξουμε το δεύτερο φάκελο που έχει σχέση με την ε, κατάληψη του άνθρακα και την ε, αναχέτηση των αρνητικών κλιματικών επιπτώσεων πρόκειται για τα μη, ρηπογόνα αυτοκίνητα. Στόχο έχουμε να αυξηθεί το μερίδιο της αγοράς για τα μη ρηπογόνα οχήματα στο πλαίσιο των αγορών από τις ε, αρχές. Στόχος θα είναι λοιπόν η μείωση των ε, ρήπων, των εκπομπών ρήπων, αλλά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο τομέα των μεταφορών. Η Ρουμανική Προεδρία καταβάλει προσπάθειες για την έγκριση της θέσης ε, του Συμβουλίου το συντομότερο δυνατό. Στη συνέχεια με τη δική σας στήριξη, το Κοινοβουλίο, προτείνουμε μια πολιτική ε, συμφωνία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Για, τώρα, ψηφιοποίηση είναι ένας τρόπος για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες μεταφορών με θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την μείωση τον, ε, του διοικητικού φόρτου. Στο δεύτερο τμήμα της Προεδρίας θα συζητήσουμε σε επίπεδο του Συμβουλίου τον κανονισμό για την ε, αποδοχή των στοιχείων ε, με ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να φτιαχτεί ένα ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο για αυτό το τομέα που θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα. Ψηφιοποίηση λοιπόν η Ρουμανική Προεδρία δεσμεύτηκε στις διαπραγματεύσεις για την ενιαία Ευρωπαϊκή Θηρίδα για την αυσιπλοεία. Στο τομέα λοιπόν της ναυσιπλοείας βασιζόμαστε και πάλι στην δική σας υποστήριξη ώστε να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία για αυτήν την οδηγία που με αφορά την κατάρτιση και την πιστοποίηση των πληρωμάτων των ναυτικών ε, ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός αμοιβαίας αναγνώρισης ε, πιστοποιητικών που χορηγούνται από τα κάτι μέλη και, την, ε, τα, χώρες. Επίσης, η ολοκλήρωση του δικτύου TEN T ε, μέσω της βελτίωσης των υποδομών και της χρήσης ε, της τεχνολογίας. Να αυξηθεί έτσι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η βιώσιμη κινητικότητα. Στόχος μας είναι στόχος προτεραιότητας γιατί θα ε, συζητήσουμε από σήμερα και στο εξής το θέματα αυτά ε, για τον κανονισμό που αφορά τον ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Διασύνδεσης ε, F2.0. Οι μεταφορές εδώ στην Ευρώπη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτά τα μεγάλα έργα υποδομή θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τα χρηματοδοτήσουμε. Ταυτόχρονα η Πυρουμανική Προεδρία ε, ε, σκέφτεται και την απλοποίηση των διαδικασιών εφόσον πρόκειται για χορήγηση αδειών πολεοδομίας αλλά και άλλων ε, διαδικασιών που θα πρέπει να διεκπαιρεωθούν ώστε να διευκολυνθεί ε, η ολοκλήρωση των δικτύων TEN-T. Ε, θέλουμε και το FEE TEN-T και γενικά να έχουμε πληροφόρηση για αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τις εποχικές αλλαγές ώρας, ε, είναι ένα θέμα που έχει πάρει μεγάλη ορατότητα και έχει αντίκτυπο Ε, φαίνεται ωστόσο να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω χρόνο για να γίνουν διαβουλεύσεις με τους διάφορους οικονομικούς ε, τομείς πριν να ληφθεί απόφαση για τα ε, εναλλαγή ώρας. Γι' αυτό και θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα μόνο στο δεύτερο τμήμα της Προεδρίας. Στόχος προτεραιότητας είναι να διοργανώσουμε και εκδηλώσεις στη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, διασκέψεις και συνεδριάσεις για διάφορα και ποικίλα θέματα. Που όλα αφορούν τις μεταφορές. Θα πρέπει να γίνει και ένα Συμβούλιο Υπουργών στο Βουκουρέστι στις 25, 27 ε, Μαρτίου ε, βασικό θέμα θα είναι οι μεταφορές και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Θα γίνει και μια διάσκεψη για τα διευρωπαϊκά δίκτυα με μεγάλη συμμετοχή των βασικών φορέων ε, του τομέα της μεταφοράς. 20 με 21 Μαρτίου διεθνής ε, συνδιάσκεψη θα διοργανωθεί για το θέμα της οδικής ασφάλειας θα οργανώσουμε λοιπόν όλα αυτές, όλες αυτές τις εκδηλώσεις στη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας Τώρα το Συμβούλιο Μεταφορών ε, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας θα γίνει στις 6 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Η ημερήσια διάταξη είναι πάρα πολύ πλούσια και τα θέματα που θα συζητηθούν ε, πολύ άριθμα. Η Ρουμανία αναλαμβάνει την ε, Προεδρία με μέρημνα στην συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ατζέντα. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο επικοδομητικό διάλογο με όλες τις δομές και κυρίως ε, στην υπηρεσία της συνέχειας και της παγίωσης του ευρωπαϊκού project, ώστε να η Ευρώπη να είναι πιο κοντά στους πολίτες, να ε, επικρατήσει περισσότερη συνοχή. Ελπίζω πως θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και πως θα έχουμε πολλά αποτελέσματα, όχι για μας, αλλά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και για όσους χρειάζονται ρεαλιστικές απαντήσεις σε το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ για το φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας σας, αλλά και πολύ φόρτο εργασίας βλέπουμε. Μπράβο λοιπόν για αυτές τις πρώτες σας εξαγγελίες. Ε, να περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Θα απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων εφόσον το επιθυμείτε στο τέλος. Κύριε Βάντεν Κάμπ, δύο λεπτά. Καλημέρα κύριε, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι η πρώτη φορά που η Ρουμανία αναλαμβάνει τα ενία του Συμβουλίου. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, λοιπόν, διότι η πολιτική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στη χώρα σας δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη την περίοδο που διανύουμε. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος με τον δικό σας ε, ενθουσιασμό και με την ε, πεποίθησή σας ότι το έργο σας θα στεφτεί με επιτυχία. Είπατε ότι θέλετε να είστε ένας ειλικρινής συνομιλητής ε, μεταξύ των ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι στο πακέτο για την κινητικότητα 1 τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει καταλήξει ακόμα σε θέση. Επίσης, διαπίστωσα το εξής. Δεν μιλήσατε για, τον, ε, για το χρονοδιάγραμμα. Το ε, η Ρουμανική Προεδρία μπορεί να προχωρήσει σε τριμερείς διαλόγους μόλις μέχρι τις 15 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η προεκλική περίοδος στην οποία δεν μπορούν να γίνουν τριμερείς, ε, ε διάλογοι. Έχουμε όμως ανοίξει το θέμα της θερινής και χειμερινής εδώ πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και το να γίνουν διαφορετικές κινήσεις από διαφορετικά κράτη-μέλη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Επίσης δεν είπατε τίποτα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Εκεί πρέπει να κατασκευαστούν ακόμα οδικές ή μεταφορικέ υποδομέ οι οποίε θα συνδέσουν τα Δυτικά Βαλκάνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο, τουρισμός. Εμείς ξέρετε είμαστε η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να συζητά το θέμα του τουρισμού. Είναι θέμα πολιτικής. Ε, όπως και για τη δική σας χώρα φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρει ο τουρισμός και για τη Ρουμανία. Ευχαριστούμε κύριο Σερτού. Ευχαριστώ Κυρία Υπουργέ, καταρχά να σα καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Μεταφορών. σα καλωσορίζω και εκ μέρου τη πολιτική ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την πρώτη Προεδρία τη χώρα σα. Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε στις ε, υποχρεώσει και στα καθήκοντα που έχετε αναλάβει. Μα παρουσιάσατε μια δέσμη προτεραιοτήτων που θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Ορθώ τι επιλέξατε αυτέ τι προτεραιότητε. Είναι τα θέματα που πραγματικά μπορούν και πρέπει να ολοκληρωθούν στη διάρκεια της Προεδρίας σας και γι' αυτό σας συγχαίρω για την επιλογή αυτών των προτεραιοτήτων. Γιατί είχαμε και στο παρελθόν ε, προεδρίες οι οποίες είχαν αναλάβει την ε, φιλοδοξία να επεξεργαστούν τα σημαντικά θέματα και τελικώς απέτυχαν. Εσείς βάλατε λοιπόν σωστές προτεραιότητες, λαμβανομένου υπόψη ότι θα γίνουν και ευρωεκλογές στη διάρκεια της προεδρίας σας με γενικό στόχο να προωθήσουμε την ε, ευρωπαϊκή πολιτική και ιδίω τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω εγώ να σημειώσω και να αναδείξω τρία θέματα, τρεις προτεραιότητες, ε, τις οποίες αναφέρετε και εσείς. Πρώτον, δίκτυα TNT, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ε, διασύνδεση με τα περιφερειακα κράτη, κράτη-μέλη. Και ξέρετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα ε, για τα περιφερειακά κράτη-μέλη, τα οποία δεν έχουν τη διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρειάζονται. Ξέρετε όμως ότι πλέον είναι αναγκαίο να γίνει το επόμενο βήμα αφού έχουν περάσει 6-7 χρόνια από τα TNT. Και το επόμενο βήμα, ακριβώ γιατί έχει αλλάξει ο κόσμο, είναι ε, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Υβριδικά αυτοκίνητα, ε, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στήλε φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υδροποιημένο φυσικό αέριο. Όλα αυτά πρέπει πλέον να τα εντάξουμε στα κεντρικά δίκτυα, στα δίκτυα TNT και θα πρέπει να αναλυφθεί δέσμευση αυτά να τα επεξεργαστούμε στην επόμενη θητεία. Αυτό βεβαίω ισχύει και για τις γενικές υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν και τέλος εγώ έχω δραστηριοποιηθεί ε, ώστε ε, να ε, καταργηθούν ε, και να αντιμετωπιστούν οι απάτες σε σχέση με τους ταχογράφους ε, ξέρουμε ότι και η δική σας χώρα έχει πληγεί ιδιαίτερως από αυτήν την ε, απάτη, οπότε θα ήθελα και η δική σας Προεδρία να αναλάβει σχετικέ πρωτοβουλίε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε κύριο Λούμπγεν. Ευχαριστώ και καλώ ήρθατε, Υπουργέ. Έχετε λίγο χρόνο για να καταφέρετε τίποτα, διότι το Κοινοβούλιο ουσιαστικά διακόπτει σε μισή μήνες, καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ. Δεν θα ήθελα ωστόσο να παρε... παραγωνιστεί το θέμα που μου είναι το προσφυλέστερο, ε, αυτών των οδικών μεταφορών. Πριν να γίνω ευρωβουλευτή, ε, είχα οδηγήσει φορτηγό επί χρόνια ε, και ξέρω πώ εξελίχθηκαν μεταφορέ από τη Σουηδία, τη χώρα μου, όπου η σουηδική μα εταιρεία εξοντώθηκε εντελώ από μεταφορικέ άλλων κυρίω ανατολικών χωρών με τιμές που ήταν περίπου το 1 τρίτο αυτό που μπορούσαμε να προσφέρουμε εμείς, γιατί ως σουηδική εταιρεία αυτές τις τιμές έπρεπε να πουλάμε για να μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις φορές μας και όλα τα υπόλοιπα. Και βεβαίως με κάθε απώλεια φορτηγού στη Σουηδία χάνουμε 70.000 ευρώ περίπου σε φορολογικό εισόδημα. Είναι πολλές οι εταιρείες που πτώχευσαν. Για μένα λοιπόν το θέμα του καμποτάζ ε, για το οποίο ο συγκεκριτής μας κάνει φανταστική δουλειά είναι ε, άκρος σημαντικό. Καλό είναι να έχουμε διεθνείς μεταφορές μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Όμω θα πρέπει να υπάρχει και δικαιότερο ανταγωνισμό. Δεν τον φοβάμαι εγώ τον ανταγωνισμό από οποιαδήποτε χώρα. Όμω πρέπει να είναι δίκαιο, θεμητό. Ε, όπου αυτό δεν είναι εφικτό εντό Ένωση, διότι αλλιώ ε, εξοντώνεται μια ολόκληρη αγορά σε ένα κράτο μέλο. Είστε μέλος και μπορεί να δέχεστε θέμα τον ανταγωνισμό από άλλο κράτος μέλος. Καταλαβαίνω ότι το θέμα του καμποτάζ του κυρίου Ερτούγκ δεν είναι και πολύ δημοφιλές όταν δούμε τις αποκρίσεις που έχει λάβει. Όμω ελπίζω να εργαστείτε κι εσεί υπέρ του δικαιότερου ανταγωνισμού. Διότι αυτοί που πλήττονται από την νομοθεσία αυτού του είδου είναι ακριβώ οι ίδιοι οι οδηγοί. Φορτηγατζίδε, νταλικέριδε που επί μήνε ε, ζουν στα φορτηγά του, στι καμπίνε των φορτηγών του και δεν έχουν κοινωνική ζωή. Ελπίζω λοιπόν ω Προεδρία να πετύχετε δικαιότερο ανταγωνισμό εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βουλή. Κυρία Μάισνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και από πλευρά των φιλελευθέρων θέλω να σας καλωσορίσω κυρία Υπουργέ. Εδώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, όπως υπόθηκε είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει η Ρουμανία την Προεδρία. Είναι και μια σύντομη Προεδρία ε, που μπορεί να σας δώσει και τη δυνατότητα να αναλάβετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και τις οποίες να τις φέρετε και σε πέρας. Ε, έχετε καταρτήσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και καλώς. Ε, αναφερθήκατε στις προκλήσεις ε, του Brexit. Εγώ ήμουνα χθε ε, στον τριμερή διάλογο και θέλω να σας συγχαρώ για την επιτυχή έκβαση του τριμερού διαλόγου για την ασφάλεια στην ναυτιλία και είδα ότι και στο single window ε, στην ενιαία θηρίδα της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας ε, τα πράγματα επίσης βαίνουν καλώς. Αναφερθήκατε στους ε, οδηγούς και στις καμπίνες των οδηγών αν και είναι μικρό το θέμα αυτό, ε, παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό γιατί ακριβώς μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορείτε να το ολοκληρώσετε ε, με θετικό πρόσημο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε εσείς. Θέλετε να... Ε, καταλήξετε σε συμφωνία στο Συμβούλιο για τα δικαιώματα των ε, επιβατών των τρένων. Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα χαροποιούσε πάρα πολύ τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και θα μπορούσε να, θέσει και μια, να δημιουργήσει μια θετική ατμόσφαιρα εν ώψη και των ευρωεκλογών. Θα ήταν κάτι που θα μας βοηθούσε και εμάς πάρα πολύ στον ε, προεκλογικό μας αγώνα. Ε, TNT, πολύ σημαντικό το ότι το έχετε θέσει ως προτεραιότητά σας. Ξέρετε ότι είναι στην ουσία το πυρηνικό, το, το βασικό, το κεντρικό δίκτυο των μεταφορών στην Ευρώπη. Μ' αρέσει πάρα πολύ και ο συγκεκριμένο χάρτης που μοιάζει με χάρτη μετρό που καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν ενέργειες και στην, ε, στις υποδομές και στην διασύνδεση τις πολυτρεπικές μεταφορές, τις οδικές, με τις χερσές, ε, με τις ε, πλωτές μεταφορές, πολύ σημαντικά και τα έργα στο Δούναβι και συμφωνώ και με αυτά που είπε ο συνάδελφος Έρτουκ. Και για το τέλος έχω αφήσει και ένα ερώτημα για την αλλαγή της ώρας. Εσείς είπατε ότι επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καταλήξει ακόμα σε θέση, θα το επεξεργαστείτε αυτό το θέμα στο δεύτερο τμήμα της Προεδρίας σας. Τι, σημαίνει αυτό δηλαδή. Περιμένετε να καταλήξει το Κοινοβούλιο πρώτα σε θέση για να δείτε τι θα κάνετε ή υπάρχουν προβλήματα και, και εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να καταλήξετε σε συμφωνία γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν αποκλίνους απόψεις και μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ Κυρία Υπουργέ, εκ μέρους των Πρασίνων θέλω και εγώ να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην πρώτη αυτή φορά που αναλαμβάνει η χώρα σας την ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Και χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε. Τρεις ερωτήσεις θέλω να σας θέσω. Πρώτον, οι μεταφορές είναι ο μοναδικός κλάδος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου από το 1990 έχουν αυξηθεί οι εκπομπές. Ε, και χωρίς αλλαγή δεν μπορούμε να αλλάξουμε ή να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ακούσαμε όμως ότι στη Ρουμανία το 1 τρίτο των ε, σιδηροδρόμων θα καταργηθούν. Ε, πιστεύετε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και πώς ακριβώς θα υποστηρίξει το Συμβούλιο την προτεραιότητα των σιδηροδρόμων όταν εσείς οι ίδιοι στη χώρα σας κάνετε το αντίθετο. Πώς γίνεται λοιπόν όταν καταργείτε σιδηροδρόμους στη χώρα σας ε, να στείλετε ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον, για μια φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα που θέλουμε να προωθήσουμε στο μέλλον. Αυτό που είπε και ε, επίσης θέλω να θέσω το θέμα του ποδηλατικού τουρισμού που τα τελευταία χρόνια ε, βρίσκεται σε άνοδο. Υπάρχει και η διαδρομή του Δούναβη. Εγώ την έκανα φέτος το καλοκαίρι. Ποδηλάτησα κατά μήκος του Δούναβη. Όμως Πρέπει να σας πω ότι στη δική σας χώρα υπάρχουν 50 χιλιόμετρα τα οποία είναι πάρα πολύ ε, επικίνδυνα και δεν μπορούσα να πάρω το ποδήλατό μου με το τρένο για να το, να το μεταφέρω. Θα ήταν μια καλή λύση αυτή να, μπορώ... να μπορούν οι ποδηλάτες να παίρνουν τα ποδήλατά τους πάνω στα τρένα. Γι' αυτό και εγώ θα ήθελα να σας καλέσω να δώσετε και το καλό παράδειγμα στη Ρουμανία, στη χώρα σας, να δείξετε ότι αυτό είναι δυνατόν, είναι εφικτό, ώστε να μπορεί να αποτελέσει αυτό παράδειγμα προς μίμηση και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και ο κύριο Λούντγκρεν μόλι αναφέρθηκε στο ζήτημα των φορτηγών. Εμεί έχουμε διοργανώσει εδώ ένα ε, συνέδριο και μάλιστα είχαμε και εδώ έναν Ρουμάνο Νταλικέρη ο οποίος ε, βρισκόταν 8 μήνες ε, στην Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο. 8 μήνε δεν είχε κοιμηθεί στο σπίτι του. Πληρωνόταν με 232 ευρώ το μήνα. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι δουλεία διότι το αίτημα για ίση αμοιβή, για ίση εργασία στον ίδιο χώρο χώρο πρέπει να εξασφαλιστεί. Εγώ λέω πάντοτε ότι μια Ρουμάνα νοσηλεύτρια που δουλεύει στη Γερμανία παίρνει τον ίδιο μισθό με τη Γερμανίδα συνάδελφό τη νοσηλεύτρια στη Γερμανία. Αλλά το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τον Ρουμάνο ε, οδηγό φορτηγού. Ευχαριστούμε κυρία Γιούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε υπουργέ. Εδώ είμαι. Ε, δύο είναι τα θέματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί είμαι και για το θέμα της συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων και για την ασφάλεια των οδικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά το ντοσχέ για τις συνδυασμένες μεταφορές, θυμάμαι ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε μια ανάλογη συζήτηση με τον Αυστριακό Υπουργό Μεταφορών, όπου μας είπε ότι μια από τις προτεραιότητες του που ήθελε εξπρές να την ε, ολοκληρώσει ήταν αυτό των συνδυασμένων μεταφορών. Όμω το Συμβούλιο ε, χρειάστηκε ένα ολόκληρο εξάμεινο για να βρει κάποια κοινή θέση. Εύχομαι. Ε, Μια και έχουν ξεκινήσει τριμερεί διάλογοι για τι συνδυασμένε μεταφορέ, εύχομαι να ολοκληρωθούν εντάχει και να φτάσουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό. Ακόμη και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, γιατί δεν έχουμε ένα ολόκληρο εξάμεινο στην πραγματικότητα. Το ντοσχέ των συνδυασμένων μεταφορών είναι ένα βασικό σημείο όπου θα μπορούσε να υπάρχει μια πραγματική καμπή και να υπάρξει ουσιαστική μείωση των μεταφορών που προκύπτουν από τις μεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Γνωρίζω ότι η Ρουμανική Προεδρία είναι ιδιαίτερα μαχητική. Ξέρουμε ότι έχετε την διάθεση να εργαστείτε και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο οπότε αυτό μας δίνει ελπίδε. Το ίδιο και σε ό,τι αφορά τις οδικές υποδομές. Πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή εγκρίναμε την εντολή, θα πάμε σε τριμερή διάλογο, ελπίζω και εδώ να υπάρξει η ίδια διάθεση από την πλευρά της Προεδρίας να φτάσει πολύ γρήγορα σε κάποια συμφωνία. Ε, θα πρέπει να πετύχουμε γρήγορα κάποιο αποτέλεσμα για να έχουμε και ένα θετικό μήνυμα να αποστείλουμε στους πολίτες. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πλούμ, μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητές σας. Ελπίζουμε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τις ε, πετύχετε. Απλώς εγώ από την πλευρά μου θέλω να σας πω ότι θα σας στηρίξω πλήρως από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Μιλήσατε για το πακέτο της κινητικότητας και έχω μια ερώτηση. Γιατί ε, ψηφίσατε, ουσιαστικά απήχατε από την ψηφορία στο Συμβούλιο. Ξέρετε ότι οι χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης δεν είναι στην ε, πιο δυνατή θέση σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή. Η πρόταση αυτή είναι πιο προστατευτική, ε, έχει περισσότερο τάσεις προστατευτισμού για τις χώρες που βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη. Στο Κοινοβούλιο, μάλιστα, ήμασταν αρκετά διχασμένοι και δεν μπορούσαμε να βρούμε μια κοινή θέση. Καταφέραμε λοιπόν απλώς να αποσπάσουμε ε, βελτιωμένε προϋποθέσεις και όρου για τι χώρε τη περιφέρεια τη Ευρώπη. Γιατί λοιπόν να η Ρουμανία κατά την ψηφοφορία. Και μια άλλη ερώτηση, η διευκόλυνση για τη δεσύνδεση τη Ευρώπη. Είναι μια από τι προτεραιότητέ σα. Σήμερα τέσσερα δι εγκρίθηκαν για να μεταφερθούν από την πολιτική συνοχή στο ΣΕΦ. Ε, η ερώτησή μου λοιπόν είναι ακριβώς για το ε, έμβασμα αυτό, αυτή τη μεταφορά και τα κονδύλια που γενικώ χρησιμοποιούνται. Έχουμε κάποια προβλήματα με τη χρηματοδότηση. Ποια είναι η κατάσταση στη Ρουμανία σε σχέση με έργα που θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από αυτή τη διευκόλυνση, από το ΣΕΦ. Ε, στην ε, τωρινή περίοδο προγραμματισμού πώ έχουν προχωρήσει οι διαδικασίε χρηματοδότηση αυτών των έργων. Διότι στο Κοινοβούλιο γίνεται πολλή λόγο για το ότι τα χρήματα υποεκτελούνται. Ευχαριστούμε, κυρία Ρεβονταλόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ Υπουργέ. Εδώ είμαι. Να με, να με. Ευχαριστώ Υπουργέ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας. Το είπαν όλοι οι συντονιστές. Είμαστε σε μια τέτοια χρονική συγκυρία που διαφέρει κάπως από τη δική σας. Πρέπει λοιπόν για τα κείμενα, από των οποίων υπήρξε πρόταση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προφανώς και του Ευρωκοινοβουλίου, πρέπει γρήγορα να ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι με το Συμβούλιο. Μεταξύ των κειμένων αυτών, των προτάσεων αυτών, υπάρχει ένα που το θίξατε στην ομιλία σας, η Ευρωβινιέτα. Αυτό που ονομάσαμε ευρωτέλο. Η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο εδώ ήταν πολύ ξεκάθαρη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την πρόταση αυτή, αλλά δυστυχώ ο κατάλογο πενταετήτων του Συμβουλίου προβλέπει η Κορεπέρ τον Ιούνιο. Ξέρετε ότι για μα ο Ιούνιο είναι ε, εκτό προγράμματο. Είναι ένα κείμενο που δεν υπάρχουν ιδιαίτερε δυσκολίε ή δυσχέρειε. Θα ήταν λοιπόν νομίζω σημαντικό για να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να προχωρούμε, να επιταχύναμε να επιταχύναμε και να προβλεφθεί ο τριμερής διάλογος σε άλλη φάση, ώστε να δυνατόν πιο γρήγορα. Να υπάρχει τελικά μια θέση του Συμβουλίου και του Κορεπέρ και των διαφόρων υπουργών για το θέμα αυτό. Ε, εδώ και δύο χρόνια συζητιέται το θέμα της Ευρωβινιέτας, όπως και τα άλλα σχετικά κείμενα. Σας παροτρύνω λοιπόν να προχωρήσετε ταχύτερα για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Διασύνδεση, θα στηρίξετε την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου υπέρ της αμοιβαιότητας, στην πρόσβαση στην αγορά ε, σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Είναι και αυτό ένα θέμα άκρο σημαντικό για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλες τις εταιρείε και τους Ευρωπαίους ε, φορείς. Ευχαριστούμε κυρία Ρεβό. Κυρία Μπιλμπάο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Υπουργέ. Ε, Καλή επιτυχία για την Προεδρία. Έχετε φιλόδοξη ημερήσια διάταξη. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω για δύο προτεραιότητες που είναι σημαντικές για την Ένωση και όχι μόνο για τους θεσμούς. Ε, πρόκειται και το ιδέσμι για την κινητικότητα. Νομίζω πως έχουμε υποχρέωση και εγώ θα ήθελα να σας παροτρύνω να σπρώξετε αυτό το πακέτο που θα μας επιτρέψει να λύσουμε ένα σωρό προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε και και το θέμα των ε, διευρωπαϊκών δικτύων. Ε, πρόκειται για προτεραιότητες ε, που είχαμε ανέκαθεν. Ε, όμως πολλά λέμε αλλά λίγα κάνουμε και θα πρέπει να συνεχίσουμε να διατηρούμε αυτή τη γραμμή, να στηρίζουμε αυτά τα project που δίνουν προς την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Για το θέμα τη αλλαγή ώρας το Συμβούλιο ενδιαφέρεται, αλλά χθε είδαμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές και ότι δεν θα υπάρξει κανένα, μάλλον συγγνώμη, αν δεν γίνονται πια αλλαγές ωραρίου δεν θα επηρεάσει αυτό ούτε την οικονομία ούτε τίποτα άλλο ε, και θα βελτιωθεί και η υγεία των πολίτων. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, να αποφασίσουμε και κάτι να κάνουμε γιατί είναι αυτή η υπόθεση για την οποία ε, ε, συμμετείχαν στη διαβούλευση περισσότεροι Ευρωπαίοι από ποτέ, από ότι για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Θα, σας, θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω την ψήφια εμπιστοσύνη γιατί η εμπειρία μου μου λέει ότι οι πιο μικρές χώρες καταφέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα στις προεδρίες και δεύτερον γιατί εσείς δείχνετε πως είστε μια προεδρία όπου συμμετέχουν πολλές γυναίκες και αυτό είναι εγγύηση για το μέλλον και για την επίτευξη καλών και θετικών αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου και κυρία Τερπαντέλ. Καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ. Η Ρουμανική Προεδρία πρέπει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις ε, και στον τομέα των μεταφορών έχουμε πολλά θέματα προτεραιότητας, ιδιαίτερα τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να ξεκινήσουν οι τριμερείς ή έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι συνάδελφοι ήδη τα πιο σημαντικά θέματα, ωστόσο θα ήθελα να σκεφτούμε την προοπτική της, το σκεφτόμαστε από την Προεδρία, από την προοπτική της Προεδρίας. Όταν έχουμε την Προεδρία μιλάμε εξ ονόματος ε, όλων των Ευρωπαίων. Όπως μπορείτε να το διαπιστώσετε, οι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου σας στηρίζουν για να μπορέσετε να επεκτείνετε τα διευρωπαϊκά δίκτυα προς τις ε, ε, περιφερειακές ζώνες, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει τα δίκτυα να φτάνουν μέχρι την άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι έχουν ε, μεταφερθεί χρήματα από την πολιτική συνοχή στην διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης και γνωρίζουμε πως η ασφάλεια στους δρόμους είναι και αυτό πρόκληση. Στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε καταβάλει προσπάθεια για να εγγυηθούμε για ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο και ελπίζουμε πως ε, θα γίνει δεκτό ε, το πλαίσιο αυτό και θα έχουμε έτσι λιγότερα θύματα στους, ε, στους δρόμους. Επίσης, μαζί με την Πρόεδρο, ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές γυναίκες στην Προεδρία της ε, Ρουμανίας, ήθελα να τονίσω το project που ονομάζεται «Γυναίκες στις μεταφορές». Ο τομέας αυτό συχνά ε, Εκπροσωπείτε περισσότερο από τους άνδρες. Ελπίζω πως θα μας στηρίξετε στο πρόγραμμα μας αυτό. Ευχαριστώ πολύ. 8 Μαρτίου είναι η διεθνή ημέρα των ε, γυναικείων δικαιωμάτων και θα είναι μια καλή ευκαιρία για να δείξουμε ότι οι ε, γυναίκες είναι πολύ άρθμες και πολύ ε, ικανές στις μεταφορές. Θα διοργανώσουμε κάτι πως είναι να δείξουμε ότι είναι συμβατό να είσαι γυναίκα και να είσαι και στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω κυρία Υπουργέ. Εδώ κάθομαι. Ναι, μιλήσατε και εσείς για αυτό το θέμα. Ένα σημαντικό θέμα είναι η οδική ασφάλεια. Αύριο θα ξεκινήσουν οι τριμερείς ε, διάλογοι, οι σχετικοί και ε, αναφερθήκατε και στις προτεραιότητες σας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα αυτό, γιατί είμαι και εισηγήτρια και θέλω να επεκτείνουμε το πεδίο ισχύω. Και ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε ανησυχίε ω προ το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Αν και δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλε οι ανησυχίε ώστε να μην καταλήξουμε σε συμφωνία, γιατί τα περισσότερα ατυχήματα δεν γίνονται στο δίκτυο TNT, αλλά εκτό αυτού του δικτύου. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα στι συζητήσει μα. Επίση, επικέντρωση τη προσοχή μα πρέπει να είναι στου πλέον αδύναμου ε, συμμετέχοντε ε, στην κυκλοφορία, δηλαδή ποδηλάτε, πεζού, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και τρίτος τομέα που πρέπει να, να, να του δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ε, η ασφάλεια, ε, ιδίως εν ώψη και της αυτόνομης οδήγησης με την κατάλληλη σήμανση κτλ. Ελπίζω πραγματικά να στεφθούν με επιτυχία οι τριμερεί διάλογοι και να ολοκληρωθούν με ε, θετικό αποτέλεσμα γιατί ε, πραγματικά ο αριθμός ε, των νεκρών στους δρόμους της Ευρώπης εξακολουθεί να είναι υψηλός. Γι' αυτό και πρέπει νομίζω να συνεργαστούμε όλοι ε, μαζί για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Κυρία Άντερσον, ευχαριστώ. Απλώ να πω ότι χαίρομαι πολύ που σα βλέπω εδώ σήμερα και ότι υποστηρίζω πλήρω τι προτάσει σα και τι προτεραιότητε σα. Θα ήθελα να τονίσω ένα-δύο πράγματα. Πρώτον, για τα μισθωμένα οχήματα. Είμαι μια από τις για το θέμα αυτό και έχει μια ταραχώδη ιστορία από τον δοσιά αυτό στην Επιτροπή μα. Θα το γνωρίζετε. Οι ψηφοφορίε στην Ολομέλεια είχαν πολύ μικρές διαφορές για να περάσει μια ή άλλη άποψη και περάσει μια τροπολογία που ε, νομίζω ότι μα προκαλεί να ξαναδούμε όλο το κείμενο από την αρχή. Ιδίω πρέπει να δούμε τι τροπολογίε που πήγαν ω την Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα. Δεν ήταν όλε ριζοσπαστικέ ή σοσιαλιστικού περιεχομένου, όπω κάτι θα έλεγαν στο ΕΛΚ. Κάποιε ήταν ιδιαίτερα ε, ορθολογικέ και ήθελαν απλώ να ενισχύσουν την νομοθεσία. Ελπίζω λοιπόν ότι το Συμβούλιο που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει τη θέση του θα κοιτάξει πολύ προσεκτικά το θέμα. Δεύτερον, για τα δικαιώματα των ε, επιβατών σιδηροδρομικών μεταφορών. Νομίζω ότι το γνωρίζετε αυτό. Ήταν μια τεράστια νίκη για το Κοινοβούλιο, διότι καταφέραμε να κάνουμε μια πολύ εξισορροπημένη και φιλόδοξη πρόταση. Ενώσει καταναλωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο την καλωσόρισαν θερμά και κάλεσαν τη Ρουμανική Προεδρία να την προωθήσει άμεσα. Ελπίζω ότι αυτό εννοούσε και η κυρία Μάισνερ. μάλιστα, εάν δείτε τις λεπτομέρειες της πρότασης, υπάρχει ε, ακόμη και δικαιολογία για τη ρήτρα της ανατέρας βίας, θέτοντας τα συμφέροντα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών ε, ως... Ε, ευθύνη στις εταιρείε. Ε, μάλλον ε, δεν την περνάει στι εταιρείε ακόμα, αλλά στους καταναλωτέ. Πρέπει εδώ να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Όταν κάποιοι χάνουν την ανταπόκρισή του. θα πρέπει να μην χάνουν τα δικαιώματά του. Για τα δύο λοιπόν αυτά ζητήματα θα πρέπει κάτι να γίνει. Για το υπόλοιπο τη έκθεση, νομίζω ότι συνεργαζόμενοι μπορούμε να προωθήσουμε επαρκώ την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Άντερσον. Κυρία Γκραπίνη, με εσά κλείνουμε τον γύρο Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε ε, και ευχαριστώ και εσάς Υπουργέ και μετά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν. Ε, κυρία Υπουργέ, η, ε, συνα... Ε, κάνατε μια παρουσίαση πολύ διεξοδική, λεπτομερή και διαφωτιστική. Δεν το λέω επειδή είμαι και εγώ από τη Ρουμανία, αλλά γνωρίζω πολύ καλά την κυβέρνηση που τώρα έχει τα ενία στη χώρα και γνωρίζω ποιο είναι το δυναμικό τη ομάδα των κυβερνώντων. Είμαι βεβαία ότι θα λάβετε υπόψη όλες τις προτάσεις των συναδέλφων. Μην ξεχνάμε ε, και να μην έχουμε και πατές, Η Ρουμανία έχει μια προεδρία κουτσουρεμένη σε σύγκριση με τις υπόλοιπε. Ε, μειονεκτή. Γι' αυτό λοιπόν να σα θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα σε ό,τι αφορά τι υδροδρομικές μεταφορές. Γνωρίζω ότι η Ρουμανία κάποια στιγμή είχε ένα από τα πυκνότερα δίκτυα στην ε, ε, Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική. Ε, θα πρέπει αυτή τη στιγμή το σύστημα αυτό να το εξυγχρονίσουμε. Πιστεύω όμως ότι λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που θα έχετε στην διάθεσή σας, μήπως θα πρέπει να ενταχθεί το θέμα των σιδηροδρομικών μεταφορών στο θέμα τη διασύνδεση και των δικτύων των διευρωπαϊκών, τα TNT. Έπειτα για τι μεταφορέ και την αντίκτυπό του στον τουρισμό. Ένα θέμα, μια διάσταση που μα έχει διαπασχολήσει. Εάν οι μεταφορέ είναι καλέ και ασφαλεί, ο τουρισμό θα ανθίσει. Σα ευχαριστώ πολύ και κάθε επιτυχία για την Προεδρία Σα Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκραπίνη, κυρία Υπουργέ. Μπορείτε να απαντήσετε σε όλε τι ερωτήσει μαζί. σε όλα τα ντοσιέ μπορείτε να σχολιάσετε και είναι και πολλά. Βλέπω ότι ανασκουμποθήκατε, θα σας δώσω αρκετό χρόνο για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, ε, Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις ερωτήσεις που μου θέσατε. σε μένα και στην Προεδρία μας. Αυτό που εγώ καταλαβαίνω και που θα ήθελα να σας πω είναι ότι στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε από κοινού το ευρωπαϊκό εγχείρημα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών μας. Αναφερθήκατε και τονίσατε στο τι θα πρέπει να κάνουμε μαζί για να προστατεύσουμε τους πολίτες αλλά και για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας προκειμένου να επικεντρωθούμε στην βιώσιμη διασύνδεση, κινητικότητα και όλες τις άλλες πολιτικές που θα υλοποιήσουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα αλλά και την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, όπως είπα και εισηγητικά, ότι η Προεδρία μας είναι και φιλόδοξη Προεδρία αλλά και ρεαλιστική. Και είμαστε ρεαλιστές γιατί ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι λίγος. Θα πρέπει στην ουσία τις εντολές που έχουμε να τις διεκπαιρεώσουμε μέσα σε δυόμισι μήνες. Και αυτό το έχουμε λάβει υπόψη μας στην κατάρτιση των πρωτοτεραιοτήτων μας. Και γι' αυτό ανέφερα ότι θέλω να ολοκληρώσουμε τους πλέον σημαντικούς φακέλους έως τα μέσα Μαρτίου, δηλαδή στις 7 Μαρτίου. Εσείς όλοι ε, είπατε, ε, ε αναφερθήκατε στους, ε, ε, στους στόχους αυτούς και στις προτεραιότητες αυτές και είπατε ότι συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Κάμπ. Έχουμε έναν οδικό χάρτη πράγματι που θα μας καθοδηγήσει στη διάρκεια της Προεδρίας μας και σας επιβεβαιώνω λοιπόν ότι έχουμε θέσει αυτές τις 7 προτεραιότητες έως ότου λήξει η δική σας θητεία. Βεβαίως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, το γενικό πολιτικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί από τις ευρωεκλογές αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτούς τους 7 φακέλους προκειμένου να ολοκληρωθούν. Όσον αφορά το πακέτο για την κινητικότητα υπαριθμών 1, θέλω να σας πω ότι παρακολουθούμε με προσοχή τα όσα έχουν συμβεί εδώ στο Κοινοβούλιο, αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Σε επίπεδο Συμβουλίου όμως εμείς είμαστε έτοιμοι διότι έχουμε παραλάβει την εντολή από την Αυστριακή Προεδρία και είμαστε έτοιμοι για την έναρξη των διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Όμως θα θέλουμε να μάθουμε αν οι συζητήσεις που θέλετε να γίνουν θα ε, αφορούν ολόκληρο το πακέτο ή αν θέλετε, και είμαστε ευέλικτοι εμείς, αν θέλετε να ε, εισέλθουμε σε τριμερή διάλογο για τον έναν ή για τον άλλον φάκελο για τον οποίο εσείς έχετε συμφωνία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να επιδείξουμε ευελιξία για να ξεκινήσουμε ε, τον τριμερή διάλογο μαζί σας για όποια θέματα ε, αυτό είναι εφικτό. Όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, αποτελούν απολύτως προτεραιότητα για της Ρουμανικής Προεδρίας. Και κατά αυτή την έννοια θέλουμε να ε, συνενώσουμε όλες τις πρωτοβουλίες και τα εγχειρήματα που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας και των, της ε, επιχειρησιακής ε, ε λειτουργίας στις, ε, στον τομέα των μεταφορών στα Δυτικά Βαλκάνια στην, ε, στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας. Επίσης, ο κύριος Έρτουκ, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για, το ερώτημα, για τα μηνύματά σας, για τα όσα είπατε και ε, μου απευθύνατε και ένα ερώτημα. Πράγματι, το δίκτυο TNT είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρουμανική Προεδρία και αυτό διότι το δίκτυο αυτό εξασφαλίζει την διασύνδεση ολόκληρης Ευρωπαϊκής Υπήρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες, για την ασφάλειά τους και θα συνεχίσουμε βεβαίως να παρακολουθούμε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στο θέμα αυτό. Θέλουμε από κοινού με εσάς να προσδιορίσουμε τις λύσεις που θα προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της κινητικότητας. Επίσης, υποστηρίζουμε και όλες τις άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί στον τομέα των εναλλακτικών υποδομών. Όσον αφορά και πάλι το θέμα της κινητικότητας. Uh, soluțiile echilibrate de compromis care să conducă la asigurarea unei. Η προτεραιότητα τη Ρωμανική Προεδρία είναι να βρούμε συμβαστικέ λύσει που να επιτρέψουν την ε, καλύτερη λειτουργία τη ενιαία αγορά, να βελτιωθούν οι κοινωνικέ συνθήκε και οι εργασιακέ συνθήκε, όσων δουλεύουν στον τομέα αυτό. Θέλουμε περισσότερη οδική ασφάλεια και καλύτερο έλεγχο. Θα πρέπει η υλοποίηση να είναι εναρμονισμένη και να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Επίση, θα πρέπει να μπορούμε να απαλλαγούμε από το διοικητικό και γραφειοκρατικό άχθο που επιβαρύνουν τι επιχειρήσει. Ο κ. Μαρινέσκου αναφέρθηκε στην κινητικότητα επίση. Βεβαίω, εδώ ε, βρίσκομαι ως εκπρόσωπος της Προεδρίας του Συμβουλίου. Εκπροσωπώ τη Ρουμανική Προεδρία και σε ό,τι αφορά την ε, ψήφο μας στο Συμβούλιο Μεταφορών να πω ότι ήμουν ε, υπουργό ασκούσα καθήκοντα απλώς ε, για τις μεταφορές στη Ρουμανία. Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω εκ μέρους της προκατόχου μου. Τώρα, γιατί απήχαμε, διότι το τελικό κείμενο δεν ε, τα στις προσδοκίες της Ρουμανίας. Η ψήφος της Ρουμανίας δεν επηρέασε ούτως ή άλλως ε, τη γενική κατεύθυνση που πήρε η ψηφοφορία. Και βεβαίως αυτό θα επηρεάσει και τη δράση της Ρουμανικής Προεδρίας. Σας έδωσα την απάντησή μου ως ε, ασκούσα καθήκοντα ε, προσωρινά για το θέμα των μεταφορών στη Ρουμανία και όχι ως εκπρόσωπος της Ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Τώρα στην ερώτηση της κυρίας του και του κυρίου Κράμερ. Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές είναι μια προσέγγιση που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να μειωθούν οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Είναι ένα από του στόχου τη Προεδρία και γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ε, το θέμα αυτό στο ευρωπαϊκό επίπεδο να προχωρήσει. Είναι προτεραιότητα ε, και θα παραμείνει. Ελπίζουμε να καταφέρουμε μια ε, εξισορροπημένη, σωστά εξισορροπημένη συμφωνία και στο Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τους δυόμισι μήνες που μας απομένουν. Ε, όσο για την αλλαγή της ώρας, ε, την θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Έχουμε δυσκολίες σε επίπεδο Συμβουλίου. Εάν στην περίπτωση του Κοινοβουλίου βρέθηκε λύση, το πρόβλημα ήταν στο Συμβούλιο. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν να συνεννοηθούν καλύτερα μεταξύ τους, να συνεννοηθούν με τις γείτονες χώρες, να συνεννοηθούν με τον εαυτό τους. Διότι ξέρουμε καλά ότι η αλλαγή της ώρας, ιδίω το πέρασμα προς τη θερινή, επηρεάζει πολύ. Επηρεάζει τον ρυθμό των οικονομικών δραστηριοτήτων και επηρεάζει και το πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες. Κυρία Άντερσον, μιλήσατε για την πρόταση για τα μισθωμένα οχήματα. Γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι πανέτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η Ρουμανική Προεδρία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, να διοργανωθούμε ώστε να γίνει εφικτή η απόκτηση μια γενική κατεύθυνση για το θέμα αυτό και προκειμένου να ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο. Έχουμε ήδη εντοπίσει κάποια ραντεβού, κάποιες ημερομηνίε για να ξεκινήσουν οι τριμερεί διάλογοι. Βεβαίω όλα όσα μπορούμε ε, θα γίνουν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα εντός του εξαμήνου της Προεδρίας μας ή τουλάχιστον για να πετύχουμε σαφή πρόοδο σε ό,τι αφορά την προσπάθεια εξέβρεση συμφωνίας για την πρωτοβουλία αυτή. Κυρία Άντερσον, αναφέρεται για τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών. Γνωρίζετε ότι το ντοσχέ αυτό ήδη έχει συζητηθεί σε τρία εξάμενα τριών διαφορετικών προεδριών και υπήρξαν τρεις εκθέσεις πρόοδου. Εν τέλει όλα ε, σταμάτησαν και βρέθηκαν σε αδιέξοδο λόγω του Brexit. Εγώ η Δία είμαι επιβάτης. Όλοι σας είστε επιβάτες και όλοι θέλετε να διαθέτετε περισσότερα δικαιώματα και ένα ε, ενιαίο και σαφές πλαίσιο δικαιωμάτων. Είναι ζωτική σημασία το πλαίσιο αυτό κανόνων να υπάρχει. Να είναι εύληπτο, απλό, εύχριστο και κάποιο να ασχολείται με την παρακολούθηση τη υλοποίηση των κανόνων. Η Ρουμανική Προεδρία περιμένει. Περιμένει με μεγάλη υπομονησία τα πορίσματα της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα αποφασίσει ε, εν συνεχεία για το θέμα αυτό ιδίως στη δεύτερη φάση της εντολής μας. Θα πρέπει να αφήσετε και λίγο χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρώσει τη μελέτη της. Για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Λιμπεράτσκι. Όχι. Δώστε μου δύο δευτερόλεπτα. Ναι, η ερώτηση της κυρίας Γκραπίνη. τα δικαιώματα των επιβατών στι δρομικέ μεταφορέ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί στην πρώτη ανάγνωση, όμω η Ρουμανική Προεδρία θα συνεχίσει την δραστηριότητά τη για το θέμα αυτό, προσπαθώντα το δεύτερο μέρο ε, του εξαμήνου μα να πετύχει αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε κατά λεπτό τι τεχνικέ ε, πτυχέ του θέματο. Χρειαζόμαστε χρόνο. Η Ρουμανική Προεδρία ε, ελπίζει να πετύχει κάποια πρόοδο για το θέμα αυτό στο βαθμό του δυνατού. σε ό,τι αφορά τις οδικές υποδομές, τα δίκτυα μεταφορών, όπως έχουμε ήδη πει, γνωρίζουμε ότι τα δίκτυα αυτά επηρεάζουν. Επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Δεν ξεχνώ τον τουρισμό. Δεν θα τον ξεχάσω. Είναι σε άνθηση, είναι σε πλήρη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλα τα κρατημέλη. Όταν ε, μιλούμε για το Δούναβι, ας πούμε, ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή. Καταλαβαίνουμε ότι όταν έχουμε ανάγκη από, τις, από υποδομές, αυτό φέρνει θετικές παράπλευρες συνέπειες και για άλλους οικονομικούς κλάδους. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν αμελούμε την προώθηση του τουρισμού. Σε διεθνέ επίπεδο τώρα θα πρέπει οι ομορφιές και τα αξιοθέατα των κρατών μελών να προβληθούν, διότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια είναι η ομορφότερη. Άρα θα υποστηρίξουμε όλα τα σχετικά έργα και προγράμματα που ε, προβάλλουν κατά κύριο λόγο τα δικά μας ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γενικότερα τις υποδομές και την ανάπτυξη του τουρισμού. Είναι κάτι το οποίο μου είναι πολύ προσφυλές ως θέμα. Άλλη απάντηση για την Ευρωβινιέτα. Στο δεύτερο μέρος του εξαμήνου μας μόλις πάψει το Κοινοβούλιο να λειτουργεί, τότε θα ασχοληθούμε με αυτό το σχέδιο οδηγίας, διότι θέλουμε να προχωρήσει. Για να προχωρήσουμε σε συμφωνία για το θέμα. με την άδειά σας θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για τους σιδηροδρόμους διότι και πάλι φτάσαμε σε ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τη Ρουμανία και εδώ μιλώ εξ ονόματα της ρουμανικής κυβέρνησης. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψουμε χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών. Θέλουμε ίσα ίσα να ε, επισκευάσουμε το σιδηροδρομικό μας δίκτυο και να το εξυγχρονίσουμε στο σύνολό του. Ε, βάσει τον ε, πρόσφατων μελετών, των μελετών, μάλλον πρόσφατα θα ολοκληρώθηκαν, θα δούμε τι έργα πρέπει να γίνουν. Αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ένα μείζον έργο για την ε, Ρουμανία. Ένα σιδηροδρομικό ε, δίκτυο, μια γραμμή αξίας περίπου ενό δι ευρώ που θα χτιστεί και σας εγγυώμαι ότι οι ράγες, οι σιδηροδρομικές γραμμές που είναι ε, ο τρόπος μεταφοράς που ρηπαίνει λιγότερο από όλους είναι προτεραιότητα για τη Ρουμανία. Αυτό ισχύει και για την υπόλοιπη Ευρώπη βεβαίως. Τελευταία απάντηση για την οδική ασφάλεια, την ασφάλεια στις οδικές μεταφορές, ερωτήσεις των κυριών Ταπαρντέλ και Αγιούτο. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας η οδική ασφάλεια θα παραμείνει μια πρώτη προτεραιότητα. Και μετά τις προσπάθειες τη Αυστριακής προεδρία να βελτιώσει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να πετύχουμε συμφωνία με το Κοινοβούλιο και να ολοκληρωθεί η εξέταση του θέματο εγκαίρω. Η Ρουμανική Προεδρία σκοπεύει να οργανώσει τρεις γύρους του διαλόγου με το Κοινοβούλιο. Ο πρώτο μάλιστα θα λάβει χώρα αύριο κιόλα. Θέλουμε να επιλύσουμε με τρόπο ρεαλιστικό τις διάφορες αποκλήσεις απόψεων της διαφωνίας και το θέμα της υλοποίησης, το θέμα της σηματοδότησης ε, και των ορίων είναι κάτι που θα το δούμε ιδιαίτερα προσεκτικά η Ρωμανική Προεδρία θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να πετύχει με τρόπο ε, επικοδομητικό την εξέβρεση λύσεων σε όλες τις πολιτικές που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σας αυτού του τόσο σημαντικού τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Νομίζω πως θα έχουμε ευκαιρία τακτικά να έχουμε επαφές ε, λόγω των τριμερών ε, το... αλλά και με το σύνολο των υπουργών γιατί ο τομέας ε, της, των μεταφορών είναι στην τελευταία ευθεία, τελική ευθεία πριν τις εκλογές. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν ότι και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην νομοθεσία. Ε, νομοθετική μας εργασία. Είστε επανειδήν λοιπόν. Εμείς σας περιμένουμε ξανά εδώ με ανοιχτές αγκάλες. Ε, σας ευχαριστώ. Είστε επανειδήν λοιπόν. Merci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 Mes chers collègues, <coughs> le dernier point. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελευταίο σημείο. Παρουσίαση της Επιτροπής της κατεξοδότηση πράξη για τα ντρόν που χρησιμοποιούνται στην ανοιχτή κατηγορία αναβάλλεται γιατί ε, ο κ. Μαρινέσκου ε, δεν είναι εδώ, αλλά ούτε και ε, ο αρμόδιος της Επιτροπής. Γι' αυτό και το αναβάλουμε για συζήτηση στην επόμενή μας συνεδρίαση 29 Ιανουαρίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα. Σας εύχομαι λοιπόν καλό απόγευμα. Κύριε Βίμπαρ Κάμπ, γρήγορα. Και ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε που ευχαριστώ Πρόεδρε που ευελιξία. Όντως υπάρχει πρόβλημα ε, όσον αφορά τις ημερομηνίες με τον κύριο Μαρινέσκο, αλλά θέλω να ακούσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να στείλει τα πιο, τις προ, πιο προς, τα πιο πρόσφατα κείμενα ώστε να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε την Τρίτη ή την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζετε, ο κύριος Ζωμαρινέσκου μπορεί να διαβάσει και να μελετήσει πολύ, σύντομα, πολύ γρήγορα. Το επέδειξε και με την επεξεργασία των τροπολογιών για το πακέτο κινητικότητας 1. Ε, Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούσε να μας ενημερώσει. Μάλιστα κύριε Βαντερικάμ, θα το στείλουμε ένα mail στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μας στείλει το σύνολο των κειμένων για να το συζητήσουμε στις 29. Πέρα συνεδρίασης.